Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Λέει και στα γαλλικά ο πρόεδρος. Να αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Σταματήστε τα πηγαδάκια. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αχα. Με ιδιαίτερη χαρά Αναλαμβάνω την Προεδρία σήμερα, μια από ο κύριο Λάινε είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Βαρκελόνη. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Είσαστε εντάξει από μετάφραση, ρωτά ο πρόεδρο. Λοιπόν, ημερήσια διάταξη. Έχετε σχόλια για την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ωραία, θεωρείται εγκεκριμένη. Ανακοινώσει του Πρόεδρου τώρα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε μία ακρόαση για τη Βαλτική θάλασσα στις 3 το μεσημέρι. Το εργαστήριο για τις κλιματικές αλλαγές και η μείωση εκπομπών πλήν του διοξιδίου του άνθρακος θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 4 με 6 και 30 το απόγευμα. Α3Ε2 είναι η αίθουσα. Ο κύριος Ζήμπα και ο κύριος Σκυλακάκης είναι που ηγούνται. Τι άλλο, πρακτικά έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της 12ης Μαΐου. Αν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνεται. Ψηφοφορία τώρα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ πολύ, ετοιμάστε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες. Για να ψηφίσουμε. Πρόκειται για μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Αυτή την έκθεση ψηφίζουμε λοιπόν. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για την ψηφοφορία. Είμαστε έτοιμοι. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος αριθμός 1, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 4, υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αυτή παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας 25 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια, τροπολίγη αριθμός 5, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία αριθμός 7 υπέρ. Όχι, κατά... Ναι, 7 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας προφορίες. Απορρίπτεται. Γιατί είχαμε 23 κατά, 18 υπέρ. Τροπολογία 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά σε λέξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστη τη ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συνεχίζουμε. Τροπολογία αριθμός 21. Στην παράγραφο 2. Γκαρντίνη, Γκροστέτ και Μπερλάτο. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τώρα. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, 16 κατά. Πάμε τώρα στην τροπολογία. 29 στην επόμενη σελίδα. Μάνερ. Παράγραφος 3. Τροπολογία 29 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Στην παράγραφο 3. Α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. 25 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 τώρα. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 33. Τροπολογία 33 διορθώνει ο πρόεδρος. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 33 πάντα. Δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Το Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 τώρα. Στην παράγραφο 4α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 47, τροπολογία 47, στην παράγραφο 5α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψήφισατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. «20 υπέρ, 20 κατά». Συνεπώς απορρίπτεται. Με δύο αποχές. Τροπολογία 49 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 τώρα στην παράγραφο 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58 τώρα, κατά τμήματα ψηφοφορία, σε δύο τμήματα δηλαδή. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα. τη 58 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά τμήματα. Σε δύο τμήματα είναι η τροπολογία αυτή. Πρώτο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 63 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60. Υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της προφορίας. 25 υπέρ 17 κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 56 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. αποχές. Κύριε Λάγκε, Πρόεδρε, την απορρίπτω την τροπολογία 67 γιατί η Σκιώδης ε, συγκήτρια επί τη σοφία της αποφάσισε ότι δεν έχει νόημα και δεν θα ήθελα εγώ να αντισταθώ σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν περιλαμβάνει η συμβαστική τροπολογία ένα ε, μέτρα συγκεκριμένα. Εδώ υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, αλλά δυστυχώς δεν ε, συμφωνεί η συγκήτρια για τα για φωσφορικά άλατα κλπ. Κρίμα που δεν υπάρχουν τέτοια συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εφόσον ε, και οι σκιώδη συζητητέ συμφωνούν, δεν μπορώ να κάνω τώρα τίποτα, οπότε αποσύρω την τροπολογία μου. Αυτή αριθμό 67, λέει η κυρία Ντελάγκε. Więc wycofujemy poprawkę. Αποσύρθηκε λοιπόν η τροπολογία 67. Στο μέλλον, όπως είπατε, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα είμαστε στη στρατηγική, ψηφίζουμε τη στρατηγική. Τροπολογία 68 τώρα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Εξήντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 τώρα. Υπέρ του κυρίου Φλόρενς. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 22-22. Απορρίπτεται λοιπόν. Εβδομήντα δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εβδομήντα τρία. Υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 18 κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 74 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 διακόπτει ο πρόεδρος. Τροπολογία 77. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79. Υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. 23 υπέρ, 21 ψηφι κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία λοιπόν. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 80. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Wszyscy oddali głos. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 23 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 81 τώρα, τροπολογία 81. Και 82, γιατί είναι ταυτόσιμες οι δύο αυτές τροπολογίες. Υπέρ, παρακαλώ. κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 83. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Υπέρ 84 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μεγάλη πλειοψηφία κατά. 31 ψήφοι κατά. Τροπολογία 85 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87, 88, 89 και 90 τώρα μαζί αυτές οι τροπολογίες γιατί είναι ταυτόσιμες Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενενήντα πέντε τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Τις τροπολογίες 95. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροποποιημένη γνωμοδότηση. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε το σχέδιο γνωμοδότησης με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 Το σημείο 5. Προφορική ερώτηση υπαριθμών 03 του 2011 των Γκροστέτ, Παρβάνοβα και Κάσμαν για την ολοκληρωμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του eu του AIDS. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γκροστέτ, μετά στην κυρία Παρβάνοβα και τέλος τον κύριο Κάσμαν. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση για την καταπολέμηση του ιού του AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικέ χώρες από το 2009 στο 2013. Η στρατηγική αυτή βασιζόταν σε, τρεις, σε τρία σημαντικότερα σημεία την πρόληψη, την ε, διάγνωση και ε, τον αντοπισμό των ευάλωτων ομάδων καθώς και των ε, περιφερειών που χρειάζονταν περισσότερη στήριξη. Δυστυχώ όμω, ο αριθμό τη μόλυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ποσοστά μόλυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γειτονικέ χώρε δεν μειώνονται. Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων ξέρουμε ότι το 30% των οροθετικών κατά μέσο όρο δεν έχουν τύχη διάγνωση και ότι παρουσιάζουν κίνδυνο τριπλάσιο, τρισήμιση φορές μάλλον μεγαλύτερο, να μεταδώσουν τον ιό του AIDS από το αν είχαν ε, τύχη διάγνωσης. Οι μισή οροθετικοί περίπου συνεχίζουν να λαμβάνουν ε, περίθαλψη αλλά πολύ καθυστερημένα και φτάνουν σε επίπεδα μόλυνσης από τον ιό πολύ προχωρημένα και τόσο αργά ώστε να μην είναι αποτελεσματική η περίθαλψη. Επίση, νέε μελέτε μα επιτρέπουν να επανασχεδιάσουμε τη στρατηγική για τον ε, ιό του AIDS, κατά του ιό ε, ε, του AIDS, εφόσον αποδείχθηκε ότι ένα οροθετικό, ο οποίο λαμβάνει αντιρετροϊκά φάρμακα, μετά τη διάγνωση βεβαίω, νωρίτερα από τη στιγμή της επιδείνωση τη Υγεία του έχει 96% λιγότερε πιθανότητε να μεταδώσει τον ιό σε μη μεμολισμένους συντρόφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει εδώ διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην παγκόσμια απόκριση κατά του AIDS. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό ο ρόλο πρέπει να διατηρηθεί. Να φροντίσουμε οι πρόοδοι και οι επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει να μην χαθούν, να εξυπηρετήσουν πραγματικά σε κάτι. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται στην Επιτροπή είναι το εξή Δεδομένου ότι θα πρέπει να κάνουμε διάμεση εξέταση του σχεδίου δράση. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει μια συνοπτική παρουσίαση των προόδων που έχουν επιτελεστεί ω σήμερα, συμπεριλαμβανομένων ε, τη ενσωμάτωση ε, των συστάσεων των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΗ για την διάγνωση του ιού του AIDS. Οι συστάσει αυτέ δημοσιεύτηκαν ήδη από το Δεκέμβριο του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επικαιροποιήσει την στρατηγική του ιού του AIDS, κατά του ιού του AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικέ χώρες δεδομένων των πληροφοριών αυτών, ιδίω σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την πρόσβαση σε διάγνωση και τον εντοπισμό. Επίσης, μετά την συνάντηση του 2011 της ε, υψηλή ομάδα κατά το 2 AIDS του ΟΗΕ από 15-18 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Ε, τα στοιχεία αυτά, ε, η σύνοδος μάλλον αυτή, Μα θυμίζει την 10η επέτειο από τη Γενική Συνόδο του ΙΕ κατά του u του AIDS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα προσασυντονίσει τη στρατηγική τη κατά του u του AIDS, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γειτονικέ χώρε και την ευρωπαϊκή τη ε, απόκριση διευρυμένη στο διεθνέ πλαίσιο κατά του U του AIDS. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε. Αποκινούμε τις συναδέλφους Αντώνια Παρβάνοβα και Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κροστέτ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα. Thank you very much, President. Uh, as, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως, όπως είπε ήδη η κυρία Γκροστέτ, και έθιξε τα βασικότερα ζητήματα. Εγώ απλώ να προσθέσω ότι όλοι οι αριθμοί που μας έδωσε εκ μέρου των τριών μας δείχνουν ότι υπάρχουν ανισότητες. Ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, εάν θεωρούνται ισότιμοι οι Ευρωπαίοι πολίτε ό,τι αφορά την ε, πρόληψη, διάγνωση και περίθαλψη κατά του ιού του AIDS και κατά πόσον μπορεί να ελέγξει στενότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δράση των ε, κρατών μελών και όχι μόνο να ε, καταρτίζει διακρατικά προγράμματα, διότι είναι πολύ ωραία στα λόγια τα προγράμματα αυτά, αλλά στην πράξη δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται, πώ χρηματοδοτούνται και εάν έχουν παρακολουθήσει στενά στην εκτέλεσή του τα τελικά αποτελέσματα τα κράτη-μέλη. Επίση, καθώ οι περιπτώσει μόλυνση από τον ιό του AIDS αυξάνονται, παρά τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τον καταπολεμήσει, τελικά πού φτάνουν τα όρια τη αρχή τη επικουρικότητα εδώ. Θα μπορούσε το μήνυμα αυτό να είναι και ανησυχητικό. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή Ε, στις μεταναστευτικές ροές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες οι οποίοι μπορεί να είναι και μολυσμένοι από χώρες της Αφρικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελε άλλος κάνει το λόγο για το θέμα αυτό. Εάν όχι, ας ακούσουμε τους εκπροσώπους της Επιτροπής σχετικά. Το κύριο Χιούμπερ πρώτα, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Yes, thank ε, Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή σας για την ευκαιρία να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή απόκριση στον ιό του AIDS. Νομίζω ότι η στιγμή αυτή είναι κατάλληλη, εφόσον είχαμε και την συνάντηση ψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη. Η στρατηγική θα πρέπει να συνεχίσει να υλοποιείται για 1,5 χρόνο. Έχουμε δύο ειδών πολιτικέ για να αντιδράσουμε στην πανδημία του ιού του AIDS. Η μία καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γειτονικέ χώρε και η άλλη έχει να κάνει με τη διεθνή μα απόκριση. Και οι δύο είναι αλληλένδετε βεβαίω με κοινού στόχου και στενό συντονισμό μεταξύ του. Ω προ την στρατηγική για την καταπολέμηση του ιού του AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γειτονικέ χώρε, Επικεντρωνόμαστε εδώ, όπως υπόθηκε, στην πρόσβαση στην ε, πρόληψη, δηλαδή τεστ, ε, περίθαλψη και υγειονομική ε, και υπηρεσίε υγεία μάλλον για τι πλέον ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού, για την καταπολέμηση των κινδύνων κατά τη κοινωνία των πολιτών και με τη στήριξη των κρατών μελών και των διαφόρων εταίρων ανά την Ευρώπη. Βεβαίω, εδώ θα πρέπει να βασιζόμαστε και όντω βασιζόμαστε στη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση τη κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ερχόμαστε στα συγκεκριμένα βέβαια ερωτήματα που τέθηκαν. Απέχουμε μόλις 1,5, έχουμε ξεκινήσει μόλις 1,5 χρόνο μάλλον την υλοποίηση της στατικής αυτής και θέλουμε ένα ε, συνολικό πλαίσιο ελέγχου για το σχέδιο δράσης και τη στρατηγική από τον ΑΣΕΚΕ. αυτό για να είμαστε βέβαιοι για την συμπληρωματικότητα της υποβολή υποβολής εκθέσεων και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε και για την συμβατότητα των εργαλείων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εργαλεία του ΩΣΑ. Εδώ μπορούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για ανισότητες, για τους παράνομους μετανάστες και όλα όσα θίξατε με, την, ε, με τις ερωτήσεις σας. Για την ενδιάμεση τώρα αναθεώρηση και καθώς έχουμε φτάσει 1,5 χρόνο μετά την υλοποίηση της στρατηγικής, είχαμε την πρώτη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ΟΑΣΕ για το πώς οι σχετικές μας δηλώσεις έχουν ε, υλοποιηθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταρτήσουμε πραγματικούς μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και εταίρων, μεταξύ του Think Tank για τον ιό του AIDS. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών με διάφορα φόρουμ στα οποία συμμετέχουν οι πολίτες και μπορούμε να ε, στηριχθούμε και στην διαδικτύωσή μας μεταξύ των πολιτών και των επαγγελματιών του τομέα τη υγεία, ώστε να προωθηθούν τα τεστ, οι δοκιμέ. Εδώ οι κατευθυντήριε γραμμέ για τα τεστ του ΟΣΕ είναι μια καλή βάση για τη στατικική μα και έχουμε σοβαρέ ε, συμβουλέ προ τα κράτη-μέλη για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η παροχή των τεστ ε, στα διάφορα κράτη. Τα θέματα αυτά τα συζητούμε μεταξύ των εμπειρογνωμονών του Think Tank που προανέφερα, θα τα συζητήσουμε και την προσεχή εβδομάδα και θα τα αξιολογήσει βεβαίως ε, και ο ΑΣΕ ε, κατά πόσον δηλαδή γραμμές αυτές είναι αποτελεσματικές. Για την επικαιροποίηση της ίδιας της στρατηγικής τώρα. Θεωρούμε, όπως είπα, ότι έναν χρόνο περίπου μετά την υλοποίηση της στρατηγικής οι βασικοί στόχοι βεβαίως παραμένουν έγκυροι, επιδιώξιμοι και δεν χρειάζεται πραγματικά επικαιροποίηση ακόμη. Ωστόσο, ενσωματώσαμε στη στατηγική και ιδίω στο πρόγραμμα δράση μια διαδικασία διαρκού παρακολούθηση και ενημέρωση. Όταν χρειαστεί δηλαδή επίσημη ενημέρωση των στοιχείων, η διαδικασία είναι ήδη εγκεκριμένη και θα τα συζητήσουμε βεβαίω αυτά με τα κράτη-μέλη, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους των γειτονικών χωρών και όλους τους ενδιαφερομένους συνομιλητέ μας. Όπως είπα, η πρόληψη, η πρόσβαση στη διάγνωση και τα τεστ είναι τα σημαντικότερα σημεία της στρατηγικής. ω προς τον συντονισμό μεταξύ των δύο στρατηγικών, υπάρχουν δύο στρατηγικές όπως ακούσατε που τρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο αυτές πολιτικές είναι συμπληρωματικέ. Ανάλογα με τις ανάγκες των ιδιαίτερων γεωγραφικών πραγματικοτήτων υπάρχουν προτεραιότητες στην καταστατική οι οποίες βασίζονται σε κοινούς στόχους, κοινέ δράσεις και οι διασυνδέσεις ε, αφορούν και το επίπεδο το πολιτικό αλλά και το ενδοπηρεσιακό της Επιτροπής. Εδώ εκπροσωπούμε τις διάφορες γενικές διευθύνσεις που είναι υπεύθυνε για τις διάφορες στρατηγικές. Είναι μαζί μου και οι συνάδελφοι από την Γενική Διευθύνση Ανάπτυξης. Πάντως αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές παρουσιάζονται και στην ανακοίνωση, τη δήλωση μάλλον που εκδόθηκε με αφορμή την Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου στο ΙΕΚ και θα καλυφθεί και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εδώ υπάρχει ένα κοινό στόχο στι στατικικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή στατικική, δηλαδή να υπάρξει συνολική καταπολέμηση του ιού με πρόσβαση στην, ε, στα τεστ, τι δοκιμέ και αναχέτηση τη ε, πρόοδου του ιού μέχρι το 2015. Εδώ Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για να απευθευθεί ο στιγματισμό, η διακριτική μεταχείριση και οι ανισότητε των φύλων. Σα ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει το θέμα μετά από την παρέμβαση της Επιτροπής, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι που αν μη τι άλλο την επόμενη φορά πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι πολύ γραφειοκρατικά χειριζόμαστε το θέμα. Στην ε, Ισπανία αυξάνει πάρα πολύ το AIDS μεταξύ των νέων. Και είναι πολύ ανησυχητική η αύξηση αυτή. Έχω μια αδερφή που πολύ θα ήθελα να την καλέσετε εδώ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνίζεται κατά του AIDS. Με παιδιά που έχει χάσει από αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι οι γυναίκες οι οποίες ε, ασχολούνται με την αγορά αυτή του σεξ ε, κολλάνε στο δρόμο. Και πρέπει να δούμε πώς θα προλάβουμε όχι μόνο το να κολλήσουν το AIDS, αλλά να κάνουν παιδιά πρώτα απ' όλα. Γιατί αυτά κινδυνεύουν να γεννηθούν με AIDS. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε απευθεία από κάποιον από αυτού του ανθρώπου να μα πει την ιστορία. Γιατί άλλο είναι η στρατηγική που υιοθετεί μια κυβέρνηση βασιζόμενη σε κάποια νούμερα και άλλο είναι να δούμε και να ακούσουμε του ανθρώπου που βρίσκονται στην πηγή και που έχουν κυρίω κοινωνικά προβλήματα. Προτείνω λοιπόν να αφιερώσουμε μία συνεδρίαση σε αυτό το θέμα. Έτσι καλώς βέβαια σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή που υποβάλλουμε γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος του κύριο Σάπταλτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oui, merci, le Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ανήκω περισσότερο στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, οπότε δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση να δώσω στον όλο προβληματισμό των βουλευτών που έθεσαν το ερώτημα, ιδίω τα όσα είπε η κυρία Κουτιέρε. Απλώ ο μόνο συσχετισμό που μπορώ να κάνω με την καθημερινή μου εργασία, την ε, στήριξη προ τι αναπτυσσόμενε χώρε δηλαδή, όπου υπάρχουν παρόμοιοι προβληματισμοί, το πώ διασυνδέεται η γραφειοκρατική λειτουργία σε επίπεδο πολιτικών φορέων και η καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούμε να παραμείνουμε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα κοντά με τους συνομιλητές μας από την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι καθημερινά μας θυμίζουν την ε, πραγματικότητα του AIDS με προβλήματα πρόσβασης στην περίθαλψη όσο και στις υπηρεσίες πρόληψης. Λίγο πολύ αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε κύριε Σαπτάλ. Η κυρία Γκροστέτ και πάλι. Με συγχωρείτε που δευτερολογώ, αλλά η μαρτυρία της ε, συναδέλφου, της κυρίας Γκουτιέρες, βρίσκω ότι είναι πραγματικά σημαντική. Ακόμη και αν είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί στον τομέα αυτό, Διαρκώς περιοριζόμαστε από τις δυσκολίες της επικουρικότητας. Πρέπει να περνάμε κάθε φορά από τις δράσεις που υλοποιούν τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν κάπως την αίσθηση ότι το ζήτημα αυτό, παρόλο που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε εδώ και χρόνια, τελικά κάπως ε, έχουμε αποθαρρυνθεί. Έχουμε χάσει την όθησή μας και δεν είμαστε σε αρκετή επιφυλακή. Υπάρχει ανάγκη καθημερινού αγώνα κατά της ασθένειας αυτής. Την ερώτηση την έθεσε μόλις προλίγου ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έθιξε μάλλον το ζήτημα μιλώντας για τους μετανάστες. Ε, οι μετανάστες που είναι πολύ άριθμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφεύγουν από τους ελέγχους στην ουσία. Από την διάγνωση άρα και την περίθαλψη. Εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μόλυνσης. Άρα δεν θα έπρεπε να, να προβλεφθούν ειδικέ συστάσεις προς τα κατημέλη για τους μετανάστες. Αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Χίμπελ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι Σημαντικά ζητήματα όλα αυτά. Πώ θα παραμείνουμε κοντά στην κοινωνία των πολιτών, λόγω χάρη. Το ανέφερα πολύ σύντομα ότι υπάρχουν φόρουμ όπου συμμετέχουν οι πολίτε, εντό των περιορισμένων μέσων βεβαίω των υγειονομικών πολιτικών. Έχουμε προσπαθήσει να κινητοποιήσουμε δίκτυα και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με ζητήματα του ιού του AIDS και σε σχέση με όσα είπε και ο συνάδελφος, πρέπει να παραμένουμε εντός πραγματικότητας. Αυτό είναι σημείο κλειδί στα πλαίσια της όλης μας στρατηγικής. Τώρα οι μετανάστες, το ζήτημα των μεταναστών, αυτό καλύπτεται σε σχέση με τι κατευθυντήριες γραμμέ του ΑΣΕ για τι ε, πλέον βάλατες ομάδε. Ο ΑΣΕ επίση έχει αναλάβει και ειδικό έργο σε σχέση με την μετανάστευση και τα ζητήματα υγεία. Υπάρχουν και άλλε ειδικέ συστάσει προ τα κρατη είναι πάντω ένα θέμα που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το συνεξετάζουμε με τα κρατημέλη προφανώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελε κανείς να πάρει το λόγο. Εάν όχι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περνάμε στο επόμενο σημείο. Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Α, przepraszam. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο 6 για την ώρα. στο υπαριθμό 6. Πρόκειται για προφορική ερώτηση της Όσα Βέστλοντ σχετικά με την παρουσία διοξίνης σε αλληλευτικά προϊόντα Φιλανδίας και Σουηδίας. Βέστλουντ. Κύριε Βέστλουντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Όπως και όλοι εδώ στην Επιτροπή μας γνωρίζουμε ότι η διοξίνη είναι από τις πιο τοξικές ουσίες που απαντώνται στο περιβάλλον. Και γι' αυτό υπάρχουν κανόνες της βενίας ε, αγοράς για την αποφυγή της τοξίνης αυτής. Ωστόσο, Φιλανδία και Σουηδία θέλουν να συνεχίσουν να πολλούν στη βάση μιας εξαίρεσης τέτοια ψάρια στους καταναλωτές. Η εξαίρεση που είχε δοθεί τότε είχε δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ότι υπάρχει κίνδυνος εάν προβούν σε υπερβολική κατανάλωση των ψαριών αυτών. Επίσης είχε απαγορευτεί η εξαγωγή τους. Οι πληροφορίες που έχουμε τώρα από τις ε, αρχές ε, προστασία καταναλωτών, τις σουηδικές δηλαδή, είναι ότι οι πληροφορίες αυτές δεν φτάνουν στους καταναλωτές. Πολλοί ε, καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τα έμβρια, για παράδειγμα, εάν οι έγκυες μητέρες, οι έγκυες γυναίκες μάλλον, ε, καταναλώνουν περισσότερα από τα ψάρια αυτά και χρειάζεται και τακτικός έλεγχος ετησίως και μόνο 7% οικογενειών με παιδιά γνωρίζουν ότι οι κανόνες αυτοί αφορούν και την Βαλτική και τη ρέγκα της Βαλτικής. Ένα ψάρι το οποίο καταναλώνουν πολύ στην ε, Σκανδιναβική Χερσόνησο σε μεγάλες ποσότητες. Και οι αρχές λένε ότι εάν συνεχιστεί η τάση αυτή θα είναι υπερβολική η κατανάλωση διοξίνης από εγγύους και από ε, μικρά παιδιά. Δυστυχώς οι Σουηδικές Αρχές δεν ανταποκρίνονται και διορωτώ τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση αυτή. Πώς θα αντιδράσει στο γεγονός ότι κυκλοφορεί τόσο πολύ διοξίδι στις Ρέγγες, στη Βαλτική θάλασσα δηλαδή, ώστε δεν επιτρέπεται κανείς να καταναλώσει Ρέγγες παραπάνω από τρεις φορές τον χρόνο. Τι κάνει εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ώστε σύμφωνα με το άρθρο που έχω εδώ και σας δείχνω αρχίζουν τώρα και τα εισάγουν οι Γάλλοι και τα σερβίρουν σε γαλλικά εστιατόρια τα ψάρια αυτά. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό αφορά μονάχα ένα είδος ρέγκας, τη λεγόμενη ξινή ρέγκα η fermented herring, αλλά για τη λεγόμενη αυτή ρέγγα η fermented herring στα αγγλικά, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν ότι έγκυες γυναίκες ή μικρά παιδιά καταναλώνουν πολλά από τα ψάρια αυτά. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν κανόνες και για τα υπόλοιπα είδη ρέγκας. Ίσως λοιπόν μπορεί να επιβληθεί μια να επιβληθεί ε, να υπάρξει μάλλον μια εξαίρεση για την ξινή ρέγγα που δεν είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος, αλλά πρέπει να ρυθμιστούν διαφορετικά τα των υπόλοιπων ψαριών που έχουν διοξίνη. Σα ευχαριστώ πολύ. Α ακούσουμε τώρα τις, ε, τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε βεβαίως και συναδέλφους που ζητούν το λόγο, η κυρία Ροτ Πέρεντ. προσπαθώ να προσελκύσω την προσοχή σας για να δηλώσω ότι θέλω να μιλήσω, αλλά βέβαια προτιμώ να ακούσω πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος, για... σηκώστε παρακαλώ τα χέρια σας. Σηκώστε τα χαρτάκια με το όνομά σας για να δούμε ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Ας λάβει το λόγο τώρα ο κύριος Φλό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Για διοξίνες και PTB τα ανώτατα όρια ισχύουν από το 2002 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δοθήσεις της ιδιαίτερης κατάστασης και της υψηλής παρουσίας διοξίνης σε προϊόντα και ψάρια από τη Βαλτική θάλασσα επιβάλλουν η Σουηδία και η Φιλανδία πολύ αυστηρές πολύ αυστηρούς περισμούς έχουν ωστόσο εξαίρεση μέχρι τέλους του έτους στις εγχώριες αγορές τα ψάρια που προέρχονται από τη Βαλτική δεν ανταποκρίνονται στα ανώτατα όρια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξαίρεση αυτή δόθηκε μετά από την απόδειξη που επέφεραν οι χώρες αυτές ότι η κατανάλωση των ψαριών αυτών δεν βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Πρωτίστως πρέπει να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές για τους κινδύνους σε σχέση με τους περιορισμούς ψαριών που έρχονται από την Βαλτική. Δεύτερον, ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι ψάρια και προϊόντα ψαριών που δεν συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια δεν θα διατίθεται στις αγορές εκτός Σουηδίας και Φιλανδίας. Η διαρκής παρακολούθηση της ε, ε, παρουσίας διοξίνη και PCB στα ψάρια της Βαλτικής θάλασσας πρέπει επίσης να είναι διασφαλισμένη. Ελέγχθηκαν και μάλιστα επιτόπου οι όροι αυτοί από τους επιθεωρητές το 2005. Η δε ομάδα επιθεωρητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τηρούνται οι κανόνες και φαίνεται το σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει την έκθεση της ε, Σουηδικής Food Staff Authority Επίσης το γραφείο των κτηνιάτων επιθεωρητών δεν βρήκε ενδείξεις για κατανάλωση τέτοιων ψαριών εκτός Σουηδίας και Φιλανδίας. Ο, παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις του συστήματος παρακολούθησης. Οι αρχές των ε, δύο αυτών χωρών μελών έχουν υποβάλει ένα σχέδιο δράσεω για να καλύψουν τα κενά αυτά. Επίση, οι χώρε μέλη παρακλήθηκαν να προσέχουν ιδιαίτερα τι εισαγωγέ ψαριών από τη Βαλτική και να κάνουν του απαραίτητους ελέγχου Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν προειδοποιήσει έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με ψάρια τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά από Σουηδία και Φιλανδία. ευχηστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εξαίρεση για Σουηδία και Φιλανδία δεν σημαίνει ότι οι δύο αυτές χώρες δεν μπορούν να διαθέτουν τα ψάρια αυτά εκτός της εγχώριας αγοράς τους, αλλά πρέπει να διασφαλίζουν ώστε τα ψάρια που καταλήγουν σε ε, άλλες αγορές θα πρέπει να συμμορφώνονται στις, ε, με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μόλυνσή τους από τις ε, ουσίες που ανέφερα. Η εξαίρεση λήγει στα τέλη του έτους και παρόλο που έχει βελτιωθεί η κατάσταση, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα, διότι διοξίνη και PCB είναι πράγματα τα οποία επιμένουν. Έτσι, οι υπηρεσίε της Κομισιόν άρχισαν προέτου συζητήσεις για το τι θα γίνει από το 2014 και μετά με τη λεγόμενη ομάδα της Βαλτικής. Εξετάστηκαν διάφορες επιλογές και τελικά η συνένεση ήταν να συνεχιστεί η εξαίρεση μόνο για ορισμένα είδη άγριου βακαλάου και πάντως για ρέγγες άνω των 17 εκατοστών και υπό τις ίδιες αυστηρές διατάξεις. Στο μέλλον θα γίνουν νέες επιθεωρήσεις από το ε, Γραφείο Επιθεωρητών Κτηνιάτρων και θα ζητηθεί η συμμόρφωση με την νομοθεσία επιδιοξίνης και από τις άλλες σκανδιναφικές χώρες. Οι λύσεις που έχει επιλεγεί μέχρι τώρα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών αλλά και των ψαράδων καθώς και την τήρηση των παραδόσεων ε, διατροφής. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο έχουν ζητήσει ορισμένοι συνάδελφοι. Θα σας διαβάσω τα ονόματα αμέσως τώρα. Γκλένις, πανι Μορκουνάιτε Ραντβιλ, πανι Ροντ Μπέρεν Νταγμάρα, πανι Καλ Σλέιτερ,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 κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα τοξινών στα ψάρια στη Βαλτική θάλασσα δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Στα ίδια καταλήγουν οι αρχές των χώρων αυτών ότι τα επίπεδα διοξίνης δεν είναι πρόβλημα για τους καταναλωτές στη Σουηδία. Μάλιστα έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα αυτά στην Σουηδία και το επίπεδο πρόσληψης διοξίνης δεν είναι υψηλότερο στη Σουηδία από αλλού. Οι Σουηδοί, διαπιστώνεται δηλαδή, καταναλώνουν το μισό από το συστηνόμενο καθημερινό επίπεδο διοξίνης. Μέχρι το μισό για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Σουηδία η ε, διατροφική αυτή παράδοση είναι σημαντική. Να μπορούν δηλαδή να καταναλώνουν τα ίδια αυτά ρέγκας. Αν όμως ανοίξετε, ανοίξετε το κουτί αυτό που σας ε, δείχνω εδώ μέσα στο δωμάτιο όλοι θα αρχίσετε να τρέχετε να βγείτε έξω γιατί είναι τόσο έντονη η μυρωδιά όπου κανένα παιδί δεν πρόκειται καν να το προσεγγίσει το ε, τρόφιμο αυτό. Μία φορά το χρόνο το τρώνε αυτό τα παιδιά το πολύ. Και το ερώτημα είναι τι ποσότητα καταναλώνει ο καταναλωτή από το ψάρι αυτό. Οι Σουηδοί καταναλώνουν ελάχιστες ποσότητες αυτής της ξινή ρέγγα και αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά. Άρα δεν είναι επικίνδυνο. Το ίδιο σημαντικό είναι να πω και ότι έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει εδώ ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να προβαίνουν στις επιλογές τους προσωπικά. Να μην τους επιβάλλουμε άνωθεν το τι θα πρέπει να τρώνε ή να μην τρώνε. Να τους δώσουμε βεβαίως τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό είναι ο ρόλος μας και αυτό έπραξε η Σουηδική κυβέρνηση. Οι αρχές προστασίας και ασφάλειας των τροφίμων στην Σουηδία συνεχίζουν να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στις εγγύους γυναίκες, στις μητέρες, ε, μικρών παιδιών και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν αυτές τι θα φάνε και πόσα. Το άλλο θέμα είναι το ζήτημα της εξαγωγής. Εδώ διεξάγεται έρευνα, διεξήχθη μάλλον έρευνα, η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν ότι έχουν εξαχθεί ξινές ρέγγες σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι η Σουηδία σέβεται τους αυστηρούς περιορισμούς που ισχύουν και εν τέλει θα ήθελα να επιμείνω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να επιτρέπει την εξαίρεση αυτή. Μην λησμονείτε τις πολλές θέσεις εργασίας που θα χαθούν στον τομέα της αλίας. Είναι επίσης ιδιαίτερα αφελής η προσέγγιση που λέει ότι θα επιτρέψουμε μοναχά την κυκλοφορία της ε, ξινής ρέγγας ενώ τις υπόλοιπες θα τις απαγορεύσουμε. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και στη Φιλανδία και στις άλλες χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική και όχι μόνο στη Σουηδία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπίλτ. κυρία Γκλένις Βίλμοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα δεν μιλούμε τόσο πολύ εδώ για Ρέγκα όσο για Σολομό. Για Σολομό λοιπόν μιλούμε. Δεν γνώριζα ότι είναι παραδοσιακή διατροφική συνήθεια των Σουηδών να τρώνε μολυσμένα ψάρια. Παιδιά που θα φάνε έστω και τρεις φορές το χρόνο Σολομό, από αυτό το Σολομό δηλαδή, ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μόνο 17% των καταναλωτών γνωρίζουν τα ε, ανώτατα αυτά όρια. Πώ θα διασφαλίσετε λοιπόν ότι οι καταναλωτέ διαθέτουν τι απαραίτητε πληροφορίε, ώστε να μπορούν να προβαίνουν στι επιλογέ για του εαυτού του, αλλά και για τι οικογένειε του. και όπω έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη εδώ ε, του αυστηρού κανόνε για τη διατροφή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες είναι ικανοποιητικό ότι μόνο 17% των ανθρώπων γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές. Και καθόμαστε εδώ εμείς και συζητούμε με άνεση αν θα δώσουμε ξανά την εξαίρεση αυτή στην Φιλανδία και στην ε, Σουηδία. Ευχαριστώ. Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση υφίσταται πολύ συχνά χειραγώγηση. Καμιά φορά μάλιστα κυκλοφορούν και αθεμελίωτες πληροφορίες. Λέχθηκε προηγουμένως ότι 70% των καταναλωτών δεν γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να καταναλώνεται τα ψάρια αυτά που προέρχονται από τη Βαλτική θάλασσα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια ισορροπία. Πώς είναι δηλαδή δυνατό ε, να διαβιβάζονται αντικειμενικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Σε δύο περιπτώσεις και στη δική μου χώρα συνέβη σε κονσέρβες βακαλάου να διαπιστωθεί περιεκτικότητα σε διοξίνη υψηλότερη από την επιτρεπόμενη. Αυτό όμως συμβαίνει και σε άλλες χώρες μέλη της Ένωσης. Εγώ θα ερωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το λεγόμενο monitoring. Υπάρχουν ενδείξεις ή υπάρχουν κάποιες τάσεις σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη αύξηση της περιεκτικότητας διοξίνης σε ψάρια από τη Βαλτική θάλασσα. Σήμερα το απόγευμα προβλέπεται συζήτηση για την οικολογική κατάσταση της ε, Βαλτικής. Μπορεί ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ε, το πρόγραμμα 1069 δείχνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η μόλυνση των ψαριών της Βαλτικής είναι ιδιαίτερα υψηλή και θα, κάνει κάποια, θα λάβει κάποια μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ και εσάς. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι ενδιαφέρομαι για την διοξίνη και τα επίπεδα της στα τρόφιμα και βεβαίω και στα ηχθιάλευρα τα οποία δίνονται ω ζωοτροφέ στα ζώα. Είναι γνωστά τα πράγματα αυτά. Είναι ασφαλώς δικαίωμα τη Σουηδική κυβέρνηση να δηλητηριάζει του Σουηδού πολίτε. Ελπίζω μάλιστα η σημερινή μας συνεδρίαση να μεταδίδεται από το ε, διαδίκτυο ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι τι συζητούμε εδώ και να τα ακούσουν τα πράγματα αυτά. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει να δηλητηριαστούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτε. Έχω ορισμένε ερωτήσει. Πρώτον, πώ είναι δυνατόν ένα ξεκάθαρα δηλητηριώδε προϊόν, η διοξίνη που είναι ξεκάθαρα δηλητήριο, να βρίσκεται σε οριακή τιμή για τα ψάρια τη Βαλτική, πώ είναι δυνατόν λοιπόν να επιτρέπεται υψηλότερες τιμές σε δύο χώρες μέλη για όλα τα ψάρια και προϊόντα ψαριών, όχι μονάχα για την ξινή ρέγγα. Ας γινόταν μια εξαίρεση για την ξινή ρέγγα σε, σε κονσέρβες, αρκεί βέβαια να αναγράφεται ξεκάθαρα για να μπορούν να τα διαβάσουν έγκυες γυναίκες, μητέρες μικρών παιδιών κτλ. Αλλά η συνάδελφος από την Σουηδία αναφέρθηκε στην αφέλεια, λέει της κυρίας Βέστλουντ, που εγώ διόλου δεν συμφωνώ, δεν βρίσκω καθόλου αφελή την κυρία Βέστλουντ, όταν μίλησε και για άλλα είδη ρέγκας. Α, τότε όμως ερχόμαστε το γεγονός το εξή δηλαδή, προφανώς δεν μιλούμε μόνο για την ξινή ρέγγα, ε, fermented herring, αλλά μιλούμε και για τα άλλα ψάρια, άλλες ρέγγες ή βακαλάους, πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος. Αυτά καταναλώνονται βεβαίως και στην Σουηδία, αλλά και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Μιλούμε λοιπόν για ψάρια της Βαλτικής, που ε, περιλαμβάνουν ε, Ρέγκα, σολομό, ήδη βακαλάου. Πώς είναι δυνατόν να το σκέφτεται καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει την εξαίρεση. Αυτά είναι γελία πράγματα και πραγματικά θα πέσει ο ουρανός και θα σας πλακώσει. να σεβόμαστε τις ε, παραδόσεις, δεν έχω αντίρρηση. Αν θέλετε να τρώτε ξινές ρέγγες ή να τις θάβετε κάπου τις ρέγγες και να τις ξεθάβετε αργότερα να τις φάτε, κάνετε ό,τι θέλετε αλλά αυτό θα είναι ένα μονάχα συγκεκριμένο προϊόν. Δεν θα μπορεί να αναφέρεται σε τίποτε άλλο. Και εγώ θα αγωνιστώ κατά ιασδήποτε εξαίρεσης ή παράτασης εξαίρεσης. Και θα ρωτήσω και εσά που είστε Σουηδοί, μήπως θεωρείτε ότι είστε οι ίδια αφελείς όταν πιστεύετε ότι τα ψάρια δεν καταλήγουν στις άλλες χώρες μέλη ή θεωρείτε ότι θα πρέπει και εμεί στι υπόλοιπε χώρε μέλη, για παράδειγμα στη Γαλλία, θα πρέπει να καταναλώνουμε δηλητηριασμένο σολομό. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό αυτό. Και εν προκειμένου είναι ανεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το πω εγώ, θα το φωνάξω προ πάσαν κατεύθυνση. Ο ΦΑΟ το 2005, όπω είπατε, έκανε μια έρευνα. Μετά από το 2005 όμω που είπατε, ξανά έκανε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν ξαναπήγε ε, επιθεώρηση του ΦΑΟ. Είπατε και κάτι που στα αγγλικά ωραία ηχεί και στα γερμανικά ίσως ακόμα καλύτερα ελλείψεις παρατηρήθηκαν στο σύστημα ελέγχου. Έτσι είπατε. Άρα δεν λειτουργεί το σύστημα ελέγχου. Το λέτε πολύ διπλωματικά, αλλά είναι σαφές ότι είδατε ότι πραγματικά μολυσμένα ψάρια από τη Σουηδία και τη Φιλανδία εξήχθησαν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω το έχει γίνει αυτό. Πώ είναι δυνατόν ελεγχθεί. Δεν είναι δυνατόν ελεγχθεί. Πόσου ανθρώπου θα βάλετε εκεί να ελέγχουν. Αυτά είναι απολύτως απαράδεκτα πράγματα. Και δεν μιλούμε εδώ για μια μικρή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενός ζυζανιοκτώνου για παράδειγμα. Μιλούμε για διοξίνη που είναι πολύ ενεργός δηλητηριώδης τοξική ουσία. Εάν το καταναλώσετε έστω και δύο ή τρεις φορές τον χρόνο σε υψηλή περιεκτικότητα προκαλεί βαρύ, βαρύτατες ζημιές σε μικρά παιδιά, σε μωρά, σε εγγύους. Είναι και καρκινογόνος. Όλοι τα γνωρίζουν αυτά. Τι καθόμαστε και συζητούμε εδώ. Πραγματικά μου προκαλεί αγανάκτηση ακόμα και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται ότι θέλει να κάνει μια ομάδα εργασίας τη Βαλτική, η οποία θα, τι θα συζητήσει, ότι ο καθένας μπορεί να δηλητηριάζει του πολίτε του όπως θέλει. Εάν κάνετε πολιτική οπορτουνιστική, πέστε το τότε καθαρά και να το πούμε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. άμα οι άνθρωποι πιστεύουν έτσι κι αλλιώ ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση την οικονομική κρίση, θα πιστέψουν ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια άλλη κρίση. Ούτε τη διοξίνη, ούτε τίποτε. Αυτή η εξαίρεση, η οποία ούτω ή άλλω είναι ένα έσχο, πρέπει να σταματήσει. Α βάλετε, α επιτρέψετε μια εξαίρεση για αυτή την υπόθεση τη ξινή ρέγγα, αλλά εκεί τελείωσε. Τίποτε άλλο. Μάλιστα σας ευχαριστώ κύριε Ροτ Προς τους Σουηδούς θα θέλατε να, να, να απαντήσετε, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, αισθάνομαι πραγματικά σοκ από αυτά τα λαϊκιστικά επιχειρήματα που προβάλλουν ε, σοσιαλιστές, αυτά τα τρομακτικά σκιάχτρα που σηκώνουν ότι δήθεν η Σουηδική κυβέρνηση αποπειράται να δηλητηριάσει τους Σουηδούς. Υπάρχει συνένεση του, στην Σουηδία ότι θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για την ε, ε Η Σουηδία είναι δημοκρατική χώρα και ο κόσμος συμφωνεί. Ταυτόχρονα ο σουηδικός λαός είναι από τους πιο ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά και επιθυμούν να μειωθούν τα επίπεδα διοξίνης, να καταναλώνουν πιο υγιή τρόφιμα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για θέματα περιβάλλοντος, αλλά θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να έχουν μια εξαίρεση για την ξινή ρέγγα τους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και πάλι. Ο λόγος του κυρίου Σλίτερ. Eh. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο είναι περίεργο είναι να ακούμε την Γόνα Μπίλτ ότι είναι αφελής η κυρία Βέστοντ. Όμως πρέπει να βασιζόμαστε στην επιστήμη. Πρέπει να βαζόμαστε στις εκθέσεις του επιστημονικού σουηδικού οργανισμού. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ των οικογενειών με παιδιά στη Σουηδία. Πρέπει να ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο καταναλώνουν ρέγγα 12 φορές το χρόνο. Συγγνώμη, 24 φορές ε, το χρόνο, διορθώνω μιλητής. Δηλαδή 12 φορές παραπάνω από ό,τι θεωρείται ασφαλές για την υγεία. Τοπική ρέγγα. Δεν είναι λαϊκισμός, δεν είναι αφέλεια να πούμε ότι είναι κακό για την υγεία. Φυσικά και είναι κακό για την υγεία. Φυσικά και δημιουργεί δυσκολίες. Είναι αφέλεια, το να παίρνει κανείς την υγεία του στα σοβαρά. Όχι, δεν είναι αφέλεια. 87% των Σουηδών γνωρίζουν το πρόβλημα της υψηλής περιεκτικότητας σε τοξίνες στα ψάρια. Όμως οικογένειες με παιδιά έχουν τα μέσα να δράσουν, να πάρουν τις αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρουν για να προστατεύσουν την υγεία τους. 13-14% των Σουηδών μόνο μπορούν να εντοπίσουν ποιο είναι το είδος ε, των ψαριών που πρέπει να αποφεύγουν για να περιορίσουν το ποσοστό τοξινών στη διατροφή τους. Είναι άρα λοιπόν δύσκολο. Άρα λοιπόν οι ισχυρισμοί να λέμε ότι η αλία θα εξαφανιζόταν αν δεν ίσχυε πια εξαίρεση αυτή, όχι δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να δούμε τις επιστημονικές εκθέσεις και τι λένε για τις συνέπειες. Πρόκειται για 35 εκατομμύρια κορώνες. Άρα δεν πρόκειται για το σύνολο του τζίρου της Σουηδική Αλίας. 90% των ψαριών που αλλιεύονται στη Βαλτική είναι μια χαρά στο βόρειο Κολμάρ, στο ύψος της Ρήγας περίπου αλλιεύονται. Εντάξει, έπειτα εξαρτάται και από το μέγεθος της Ρέγκας. Το ίδιο ισχύει και με τους Σολομούς. Άρα λοιπόν οικονομικά μιλάμε για μια μικρή τάξη μεγέθους. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία. Περί αυτού πρόκειται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, κυρία Βέστιλον. Δηλαδή η εξαίρεση να διατηρηθεί μόνο για την ξένη ρέγγα. Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί το να φάω που και που, αλλά μόνο 9% των Σουηδών τρώνε πάνω από μία φορά το χρόνο αυτή την ξένη ρέγγα. 84% των οικογενειών με παιδιά δεν τρώνε ποτέ δεν το βάζουν στο σπίτι. Ούτε για τα παιδιά, ούτε για τους γονείς. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στι συνήθειες, τις τοπικές, τις διατροφικές και τις επιπτώσεις από την άλλη μεριά που έχουν αυτές στην υγεία. Αυτό που είναι καλό με την εξαίρεση είναι ότι μπορεί να διακανονιστεί το θέμα του πάνω από 17 εκατοστά. Υπάρχουν ε, ζώνες φυσικά οι οποίες εξαρτώνται οικονομικά από την αλία, ζουν από αυτήν, μπορούν να επιβιώσουν όμως γιατί με τα 35 εκατομμύρια κορώνες μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Είπαμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό. Μια τέτοια απώλεια μπορούν να γίνουν άλλα πράγματα με χρηματοδότηση εφόσον υπάρξει κάποια αποζημίωση. Νομίζω λοιπόν ότι λύσεις υπάρχουν. Πολλοί γελείς πραγματικά θα πληγούν από ένα τέτοιο μέτρο. Η Κομισιόν θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Πρόκειται για μικρά ποσά, για χαμηλά ποσά. Απ' την άλλη μεριά όμως η ζημιά στην υγεία είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε εδώ την ε, πρόταση. Ελάχιστοι άνθρωποι τρώνε πάνω από μια φορά ε, το χρόνο ξινή ρέγγα. Και έτσι κι αλλιώς θα το κάνουν όσο και αν ξέρουν ότι θα πληγεί η υγεία τους, γιατί ε, το θέλουν πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ, έχουν ε, μονιδέα. Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί στην ξινή ρέγα και μόνο η εξαίρεση αυτή. Αυτός θα ήταν ο καλός συμβιβασμός. Η κυρία Σοφικόνη τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ ανακαλύπτω μόλις τώρα αυτή την κατάσταση και ανησυχώ. Γιατί σήμερα θεωρώ ότι ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τι καταναλώνει και πρέπει να ξέρει τι περιλαμβάνουν τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος και όσο γίνεται καλύτερα ενημερωμένος. Και μία από τις βάσεις της Ευρώπης το κάτω-κάτω είναι η προστασία του καταναλωτή. Άρα το πρώτο είναι η πληροφόρηση. Δεύτερον, για τις διοξίνες αυτές. Θέλω να ξέρω η προέλευση ποια είναι. Είναι φυσική, δηλαδή από τα δάση, από τα ηφαίστεια, από τι. Ή πρόκειται για βιομηχανικής προέλευσης τοξίνη. Γιατί είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα στη μία και στην άλλη περίπτωση. Το να καταναλώνουμε διοξίνη γνωρίζοντας ότι προέρχεται από φυσικές πηγές είναι λιγότερο σοβαρό από την τοξίνη που έχει βιομηχανική προέλευση. Ποια είναι λοιπόν η προέλευση αυτής της τοξίνης. Δεύτερον, ήδη πρόκειται για μια οργανική ουσία η οποία δεν εξαφανίζεται εύκολα, είναι καρκινογόνος, πρόκειται για την πρώτη κατηγορία και μένει στον ανθρώπινο ιστό για 8 χρόνια. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αν λοιπόν πρόκειται για μια συνήθεια να καταναλώνουν οι άνθρωποι εκεί αυτή την ξινή ρέγγα η οποία περιλαμβάνει διοξίνη σε μερικές χώρες συμβαίνει ωραία και δεν έχω πρόβλημα εφόσον οι καταναλωτές είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Όμως θα ήθελα να υπάρξει πραγματικά έλεγχος στις εξαγωγές. Εγώ στη Γαλλία δεν ε, νομίζω ότι θα μας άρεσε να καταναλώνουμε ψάρια που περιλαμβάνουν ένα ποσοστό διοξίνης. Δεν έχουμε εμεί τέτοια συνήθεια. Οπότε δεν θα ήθελα τέτοια ψάρια να εξάγονται και να φτάνουν στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες μέλη αν δεν το γνωρίζουμε και δεν έχουμε αποφασίσει να το δεχτούμε. Άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένη ενημέρωση για τα προϊόντα αυτά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είμαι υπέρ της αρχής της πρόληψης για να προστατεύονται οι πολίτες, αλλά είμαι και υπέρ της αρχής της προφύλαξης απέναντι στη βιομηχανία. Είδαμε τι έγινε με το ισπανικό αγκουράκι. Είδαμε πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση μετά για, την, ε, για τον κλάδο των οποροκυπευτικών της Ισπανίας. Άρα λοιπόν, ναι, ενημέρωση, αλλά προηγουμένω να γίνονται μελέτες. Υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν ειδικοί υπάρχει επιστημονική έρευνα. Πρώτα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη έρευνα και μετά η ενημέρωση για να μην δημιουργούμε προβλήματα σε μια οικονομική δραστηριότητα για λόγους οι οποίοι τελικά δεν ισχύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Κόνη. Η κυρία Σάτο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. κάτι το οποίο η Φιλανδία και η Σουηδία δεν το λένε πολύ τώρα που θέλουν να έχουν την εξαίρεση είναι ότι είναι είδος προς εξαφάνιση ο άγριος ολομός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υποθεί. Αν λοιπόν η περιεκτικότητα διοξίνης στα ψάρια είναι απαράδεκτη, και το είδος είναι υπό εξαφάνιση, τι νόημα έχει να δεχόμαστε μια τέτοια εξαίρεση για αυτό το ψάρι και να αφήνουμε να πωλείται ελεύθερα για ανθρώπινη κατανάλωση. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη συζήτηση που γινόταν στη χώρα μου, στη Φιλανδία, τότε που αγωνιζόταν για την εξέρεση, να πετύχει την εξαίρεση αυτή η Φιλανδία. Πρέπει να σας πω ότι όσα υπόθηκαν τότε δεν ήταν όλα πραγματικότητα. Διάφορες δικαιολογίες, προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν, οι όροι ήταν οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι. Βάσει όμως πρόσφατων μελετών φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν είναι καλά ενημερωμένοι ή εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται. Συνεπώς, οι, μόνο οι πιο ηλικιωμένε γυναίκες γνωρίζουν τα προβλήματα της κατανάλωσης ε, ρέγκας ή σολομού από μία ποσότητα και πάνω. Οι πιο νέες γενιές δεν το γνωρίζουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν το γνωρίζουν. Ούτε οι νέες μητέρες, ε, οι έγκυες κλπ. Συνεπώς, το σύστημα ενημέρωσης δεν λειτουργεί τόσο καλά. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ιδιαίτερα οι πιο νέοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Ένα άλλο θέμα Μια άλλη εξήγηση, τότε που θέλαμε την ε, εξαίρεση αυτή, ήταν ε, ότι η ξενή ρέγγα είναι φτηνή. Είναι για καθημερινή κατανάλωση. και ότι περιλαμβάνει και συστατικά που είναι πολύ χρήσιμα για την ανθρώπινη υγεία. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν ευαίσθητη υγεία Αν δεν υπάρχει πια αυτή η εξαίρεση, θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλες λύσεις λιγότερο υγιεινές. Αυτό μπορεί να ισχύει για την ε, Βαλτική Ρέγκα, δεν ισχύει όμως για το Σολομό. Γιατί ο Σολομός πριν από 100 χρόνια μπορεί να ήταν ε, καθημερινή τροφή γιατί ήταν ε, ευθυνός αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το Σολομό για να τον έχουν καθημερινά στο τραπέζι τους. Άρα δεν ισχύει. Αν δηλαδή βγάλουν από τη διατροφή τους οι άνθρωποι τον ε, Σολομό αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναγκαστούν να διαλέξουν λιγότερο υγιεινές αναλλακτικές λύσεις. Συνεπώς, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει ορθολογική εξήγηση για να συνεχίσει η εξαίρεση με την μορφή που είναι σήμερα. Επίσης, την Φιλανδία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λιγότερες διοξίνες στις μικρές ρέγγες της Βαλτικής. Οπότε, το πρόβλημα είναι τα πιο μεγάλα ψάρια και σε μέγεθος και σε ηλικία. Οπότε αν βγει ο Άγριος Σολομός από την εξαίρεση αυτή και αν βάλουμε ένα όριο μεγέθους για τη βαλτική ρέγγα, αυτό λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα που συζητάμε. Και η μεγαλύτερη βαλτική ρέγα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται μόνο σε κονσέρβες. Με βέβαια προειδοποίηση απάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σατοχάση. Ας διαβάσω πάλι τον κατάλογο ομιλητών. Καρλ ε, Χάινς Φλόρενς, Παν Κρίστοφ Φιέλνερ, Χορτ Σνέλχαρτ, Κρίτον Αρσένιστ, Πάνι Λίντα Μακέδεν και Πάνι Ασαβέστρου. Ε, teraz w kolejności Marit Polsen. Η κυρία Πόλσεν πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευθύ εξ αρχή λέω ότι αναγνωρίζω ότι είμαι υπεύθυνη για την εξαίρεση αυτή που πριν από 10 χρόνια πέτυχε η Σουηδία. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Βέσλουντ και με την ε, κυρία Ροτ Μπέρεντ για τις διοξίνες. Η πρώτη εξαίρεση ήταν ξεκάθαρη. Μιλούσε για απαγόρευση εξαγωγών. Συνεπώς, δεν πρέπει να μεταφέρονται οι ουσίες αυτές ούτε με εξαγωγές ούτε και μέσω ζωοτροφών. Η εξαίρεση αυτή λοιπόν θα μπορούσε να παραταθεί για λόγους πολιτιστικούς κύρια. Διότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ξινή ρέγγα στο κεντρικό Νόρλαντ όπου και καταναλώνεται περισσότερο και αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, της Βαλτικής. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προϊόντα που καταναλώνονται και προέρχονται από, την, ε, από τα προϊόντα αυτά. Πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχυθεί, να είμαστε δηλαδή πιο αυστηροί όσον αφορά τις προδιαγραφές ενημέρωσης. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που φτάνει τελικά στο κοινό. Γιατί πάνω απ' όλα πρόκειται για το τι είδους μήνυμα ε, αντιλαμβάνονται και αφομοιώνουν οι άνθρωποι ναι μεν στην εξαίρεση, αλλά ενίσχυση της ενημέρωσης των επισημάνσεων που έχουμε στις ετικέτες των προϊόντων. Η υποχρέωση επίσης μεγαλύτερου ελέγχου όταν πρόκειται για τις ετικέτες. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εξαίρεση, οι κανόνες πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί. Γιατί υπάρχουν τώρα τόσο πολλέ διοξίνε στη Βόρεια Βαλτική, είτε πρόκειται για τη Φιλανδία, είτε πρόκειται για τη Σουηδία. Πρόκειται κυρίως για τον χαρτοπολτό, πρόκειται για τη βιομηχανία χάρτου, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτέ. Πριν από 100 χρόνια, όχι σήμερα, πριν από χρόνια όμως, έβγαιναν διοξίνες και ξέρετε ότι η βιομηχανία αυτή είναι τεράστια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε λιγότερη διοξίνη, πολύ λιγότερη και μειώνεται έτσι κι αλλιώς ε, συνεχώς. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν νέες πηγές μόλυνσης με PSB με διοξίνη στην περιοχή. Στη συνέχεια, το ποσοστό διοξίνης στο μητρικό γάλα επίσης μειώνεται κατά 6% το χρόνο στη Σουηδία. Δεν λέω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε όπως και πριν, αλλά αν μη τι άλλο λέω ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την πηγή μόλυνσης. Οι κανόνες όμως πρέπει να είναι πιο αυστηροί όπως είπα. Οι ετικέτες ε, πρέπει να προσέχουμε τι αναφέρουν, να είμαστε πιο αυστηροί και σε αυτό. Να ξέρουμε αν πρόκειται για την ξινή ρέγγα ή όχι. Πάντως τα, το ψάρι αυτό δεν θα πρέπει να μεταπείτε. Η ξινή ρέγα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε επίσης σε άλλα ε, φαγητά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν για παράδειγμα κεφτεδάκια από ψάρι ε, στις ζωτροφές να χρησιμοποιείται το προϊόν αυτό. Και αυτό για να έχουμε ένα συμβιβασμό, ο οποίο να λειτουργεί καλά, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο. Η ζωή πάντα είναι περισσότερο γκρι παρά άσπρη μαύρη. Άρα δικιά μας αποστολή, κύρια αποστολή δικιά μας είναι να πετύχουμε ένα συμβιβασμό για να σεβαστούμε τις πολιτιστικές συνήθειες αλλά και για να μειώσουμε το ποσοστό δηλητηρίου που περιλαμβάνεται στα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πόλσεν. Η Φρανσουάς Γκροστέτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, άκουσα τους ε, συναδέλφους που έρχονται από χώρες της Βαλτικής. Εδώ όμως βρισκόμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, όχι εσωτερικής αγοράς, έτσι. Αυτή είναι ακριβώς και η διαφορά. Εδώ ε, οφείλουμε να, να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και της υγείας του μέσω της δράσης της Επιτροπής μας. Οι συνάδελφοι λοιπόν ας καταλάβουν και τις δικές μας τις απορίες. Καταλαβαίνουμε μεν, συνειδητοποιούμε ότι για κάποιους τοπικούς πληθυσμούς οι παραδόσεις είναι σημαντικές. Κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του. Και εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω συγκεκριμένα τη Σουηδία ή τη Φινλανδία, γιατί σε κάθε κράτος μέλος μπορεί κανείς να βρει τέτοια θέματα παρόμοια. Όλους μας αγγίζουν τέτοιου είδους προβληματισμοί. Όμως νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία να υπάρχει η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση του καταναλωτή. Εγώ δυσκολεύομαι ακόμη και να θέλω να καταλάβω τα επιχειρήματα των συναδέλφων. Πώς να δεχτεί κανείς ότι μπορεί να υπάρχει εξαίρεση εδώ. Υπάρχει διοξίνη, μιλάμε για προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία και παρόλα αυτά δεχόμαστε την κατανάλωσή τους. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει και δεν καταλαβαίνω τα επιχειρήματα κάποιων συναδέλφων. Υπό τους όρους αυτούς, νομίζω, σημαντικό είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όμως αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι σε καλά επίπεδα πλέον. Είχαμε τις διοξίνες, το βακτηρίδιο που τόσο πολύ έχει συζητηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Διαρκώς αντιμετωπίζουμε κρίσεις διατροφικές, ζητήματα ασφάλειας ε, διατροφικής και υγειονομικής. Δεν μπορούμε δεν μπορούμε όταν ε, πρέπει να απευθυνθούμε στους πολίτες να τους λέμε «Α, αυτή η εξαιρεσούλα μπορεί να υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει και άλλη μία αλλού όμως». Πώς να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή, κατά με, έχει καθήκον να μας δώσει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τα στοιχεία για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρέπει να ενημερώνουμε τους καταναλωτές, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έγκυους γυναίκες, με παιδιά, με ολόκληρο τον πληθυσμό. Το πρόβλημα είναι ότι λέμε σήμερα, εντάξει, ο άγριος ολομός ε, μη εκτροφής ε, μπορεί να έχει πρόβλημα. Πριν λίγο καιρό λέγαμε ο ολομός εκτροφής επίσης έχει πρόβλημα. Ε, άμα τα ακούσει κανείς όλα αυτά σήμερα, αρχίζει και διαρωτάται τι να φάει. Υπάρχει λοιπόν ε, πολλή δουλειά μπροστά μας εδώ. Στην Επιτροπή αυτή πρέπει να έχουμε απαιτήσει. Πρέπει να έχουμε απαιτήσει για τη διατροφική και επισητιστική ασφάλεια και υγεία. Είναι σημαντικό. Εξαίρεση λοιπόν, αλλά εγώ τη βρίσκω ενοχλητική. Ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτ, ο κύριος Φέλνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάει καιρός τώρα που δεν έχω συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση για ένα και μόνο προϊόν. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που τόσοι Σουηδοί συμμετέχουν σε, αυτό σε αυτή τη συζήτηση. Ίσως γιατί ακριβώς μιλάμε για την ξινή ρέγγα. Εάν το συγκρίναμε με κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι το Σαρκράουτ για την ε, ε, ε, Γερμανία, η φέτα των Ελλήνων ή το προσούτο της Ιταλίας. Τέλος πάντων, προφανώς είναι ένα σημαντικό προϊόν από άποψη πολιτιστικής παράδοσης. Γι' αυτό τόσο πολλοί ενδιαφέρονται και ανησυχούν γι' αυτό οι συνάδελφοι. Νομίζω σήμερα έγινε καλή συζήτηση, καλή συζήτηση για το επίπεδο του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω επίσης ότι αυτή η προφορική ερώτηση έχει το νόημά τη και καταλαβαίνω γιατί κάποιοι ζητούν την ε, παράταση της εξαίρεσης για την ε, ξινή Είναι ένα σημαντικό προϊόν για τη Σουηδία λοιπόν. Όμως το γεγονός ότι συζητήσαμε τόση ώρα για το θέμα αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ακόμη και αν υπάρχει μια εξαίρεση de facto για την ε, ξινή ρέγγα, αυτό δεν αρκεί. Εάν υπάρχει απλώς μία εξαίρεση θα έχουμε αρκετά ψάρια στην αγορά για να γίνει τελικά η παραγωγή της ξενής ρέγκας γιατί οι αλλοίς που εμπλέκονται σε αυτό το εμπόριο είναι αλλοίς χωρίς πολλά μέσα σε μικρές τοπικές κοινότητες δεν ασχολείται κανείς με την αλία μόνο, με την αλίευση μάλλον ενός μόνο είδους, ενός συγκεκριμένου μεγέθους για να φτιάξει αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, γίνεται αλίευση πολλών άλλων ειδών ταυτόχρονα από τους ίδιους ανθρώπους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό ότι αυτό το χαρακτηριστικό προϊόν που είναι όπως η φέτα, το προσούτο θα βρεθεί εκτός αγοράς. Η εξαίρεση αυτή λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία και φαίνεται να μην έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ως τώρα. Έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα. Οι Σουηδοί δεν έχουν υψηλότερα επίπεδα διοξίνη, ε, ούτε είναι εκτεθειμένοι περισσότερο από άλλου πληθυσμού στην Ευρώπη. Αυτό το ξέρουμε. Είναι αποδεδειγμένο. Και βεβαίω τα επίπεδα τη διοξίνη στη Βαλτική μα ε, ανησυχούν, όμω υπάρχει και μια μείωση κατά 6% το χρόνο. Ε, με την εξαίρεση λοιπόν αυτή δεν είδαμε να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα υγεία από ό,τι υπήρχε προηγουμένω. Οι περισσότεροι Σουηδοί γνωρίζουν τα προβλήματα που, δημιουργούν το προϊόν, που δημιουργεί το προϊόν αυτό και οι περισσότεροι γονείς τα γνωρίζουν, είναι ενημερωμένοι. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα της στατιστικής, ε, κατά πόσο είναι επαρκώς ενημερωμένοι όλοι. 17% λοιπόν των γονέων γνωρίζουν τα προβλήματα των προϊόντων μόνο, αλλά 40% των Σουηδών με παιδιά δεν καταναλώνουν αυτό το προϊόν και ένα άλλο 40% τα καταναλώνουν αλλά σπάνια. Λοιπόν, Καλά λέει η συνάδελφος και έχει δίκιο, δεν είμαστε πάντοτε σωστοί, δεν ακολουθούμε τα ενδεικνυόμενα επίπεδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΦΑΟ, αλλά πάλι σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ίσως να είναι 400 τα παιδιά που συνολικά δεν ακολούθησαν τα ενδεικνυόμενα επίπεδα πρόσληψης καθημερινής. Ας δούμε όμως συνολικά ε, το πρόβλημα και λίγο πιο σφαιρικά. Εδώ δεν μιλάμε για το πόσο θα, πόσο κινδυνεύουν κάποια παιδιά να δηλητηριαστούν μέσα σε μια χρονιά από διοξίνη. Αυτό το πρόβλημα σχεδόν δεν υπάρχει. Μιλάμε για την κατάργηση ενός ολόκληρου τομέα ελευτικού. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι εδώ το τοπίο πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Κάποιος έδωσε ένα παράδειγμα για την εξαγωγή 300 κιλών αυτού του ψαριού. Μα αυτό είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Δεν εξάγεται παντού στην Ευρώπη το συγκεκριμένο αυτό προϊόν από ψάρι. Δεν το τρώνε παντού στην Ευρώπη. Δεν κινδυνεύει όλο ο ευρωπαϊκό πληθυσμό να δηλητηριαστεί. Μην κάνουμε λοιπόν αντιδράσει υπερβολικέ εδώ για να αν καταργούσαμε αυτή την εξαίρεση αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα ήμασταν υπερβολικοί. Θα ήταν σαν να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, με μια πραγματικά έντονη αντίδραση. Καλύτερα να πληροφορούμε καλύτερα τους καταναλωτές και να μην αποθαρρύνουμε άλλο τους Σουηδούς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιέλνερ. Έχω και εγώ εδώ μια ερώτηση. θα μπορούσε να γίνει παραγωγή ξινής ρέγκας χωρίς διοξίνη. Είναι αυτό εφικτό ή είναι αδύνατο. Δεν γίνεται με άλλου είδους ρέγκα να παραχθεί αυτό το προϊόν επίσης. Uh, το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται ψάρι μεγάλου μεγέθους. Ρέγκα. Πρέπει να είναι μεγάλη και λιπαρή εάν τις αλλιεύσει κανείς το καλοκαίρι, έχουν ψηλότερα επίπεδα μόλυνσης. Αμέσως μετά το λιώσιμο, πριν από, από την περίοδο μετά το λιώσιμο των πάγων του χιονιού. Η διοξίνη ε, στη ρέγγα της Βαλτικής είναι συνήθως κάτω από το προβληματικό επίπεδο. Και τέλο πάντων είναι λίγοι οι καταναλωτέ που καταναλώνουν το προβληματικό προϊόν. Πάντω, εάν πείτε ότι μειώνεται το επίπεδο διοξίνη στο γάλα θυλασμού, όχι, λάθο είναι αυτό. Το, τα μπερδεύετε όλα. Τα επίπεδα PCB στην ε, ρέγκα τη Βαλτική έχουν ε, μειωθεί από το 78 και μειώνονται διαρκώ. Κατά 4-10% ετησίω. Όμω τα επίπεδα PCB και αυτά μειώνονται στα ίδια ακριβώ επίπεδα κατά ένα 4-10% το χρόνο. Όμω η διοξίνη, το PPDE που λέμε εδώ πέρα, δεν έχει σοβαρή μείωση. Όχι το PCB στο μητρικό γάλα έχει μειωθεί, αλλά όχι το PPDE. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί στα ψάρια μεταξύ του 1992 και του 2008 δεν υπάρχει σοβαρή μείωση του επίπεδου PPDE. Άρα τα επίπεδα διοξίνη ούτε στο μετρικό γάλα ούτε στα ψάρια έχουν μειωθεί. Το PCB είναι αυτό που μειώνεται ετησίω. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μην κάνουμε όμω τέτοιου αλληλού σχετισμού μεταξύ των δύο. Κύριο Φιέλνερ, ευχαριστώ πολύ. Μην περάσουμε τώρα σε διάλογο μέσα στο, στη συζήτηση. Απλώ να απαντήσω στην ερώτησή σα. Έχω ψαρέψει κι εγώ ίδιο ρέγγα στη ζωή μου. Δεν αγορεύομαι βέβαια τα αλλιεύματα αυτά. Αλλά ακριβώ όπω είπε ο συνάδελφο, μα έχει πότε αλλιεύεται το συγκεκριμένο ψάρι. Οπότε το μέγεθο ε, έχει κάποια σχέση με το επίπεδο διοξίνη. Εάν όμω κάποιο είναι ένα κλασικό ψαρά ε, που κάνει παράκτη αλεία και πρέπει να ζήσει από την αλεία και αυτού του ψαριού, πρέπει ακριβώ για να καλύψει τι ανάγκε τη αγορά να ψαρέψει το ψάρι τη σωστή στιγμή μέσα στον χρόνο. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουν να αλλιεύουν αυτό το ψάρι οι ψαράδε μα ε, τη σωστή στιγμή του χρόνου για να γίνει παραγωγή του προϊόντο αυτού πρέπει να υπάρχει εξαίρεση. Βεβαίω η Σουηδία δεν θέλει να δηλητηριάζει του πολίτε τη, αλλά Δεν måste, Ναι, έχω ένα κατάλογο εδώ και πρέπει να τον ακολουθήσουμε όμως, ε, ο Η κυρία Βέστηλον, αυτά που λέει ο Κριστόφλ είναι αλήθεια. Φυσικά και οι αλείς θέλουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, να συνεχίσουν να ψαρεύουν σολομό για παράδειγμα που είναι η κυρία πηγή των εισοδημάτων τους. Δεν πρόκειται για συγκεκριμένο μέγεθος ρέγκας για την ξινή ρέγκα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι οικονομικές συνέπειες έχει κυρίως η ελίευση του Σολομού. Μην κοροδευόμαστε. Η βιομηχανία εξαρτάται από το Σολομό κυρίως και όχι από τη ρέγκα. Πρόεδρος, να ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα. Είμαστε πράγματι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να κοιτάμε ολόκληρη την πτυχή του ζητήματος. Εδώ μιλάμε για την υγεία των καταναλωτών. Σύμφωνη. Ας κοιτάξουμε όμως λίγο παλιότερα. Ας ε, δούμε πώς έχουν τα πράγματα πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της ε, Σουηδίας. Η εξαίρεση παραχωρήθηκε γιατί ακριβώς η ενημέρωση του πληθυσμού ήταν πολύ καλή. Σε αντίθεση με τις βελτικές χώρες, τις οποίες δεν, δώσαμε, δεν παραχωρήσαμε εξαίρεση, γιατί θεωρήσαμε ότι η ενημέρωση του πληθυσμού εκεί δεν ήταν αρκετά ικανοποιητική. Συνεπώς, πώς γίνεται η πληροφόρηση αυτή. Μόνο 17% ενημερώνεται Λέτε, μα είναι δυνατόν, δώσαμε μια τέτοια εξαίρεση, κάτω δηλαδή από στραβές ε, ιδέες ή όχι. Για τη διοξίνη, πρέπει να ξέρουμε ότι η διοξίνη υπάρχει παντού στον κόσμο. Σήμερα τρώμε σαλάτα, ε, έχει διοξίνη. Βέβαια αυτό που έχει σημασία είναι ε, το ποσοστό, είναι οι ποσότητες διοξίνης που περιλαμβάνονται. Βεβαίως πάντοτε <clears throat> χρειάζεται περισκεψή. Το ερώτημα είναι όταν πρόκειται για παραδόσεις και όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και οι στατιστικές που βλέπω εδώ της εταιρεία Προστασίας της Φύσης ότι είναι, της δηλαδή, ότι είναι 6% περιέχουν διοξίνη. Ενώ πολλά από τα άλλα το υπόλοιπο ποσοστό των ψαριών δηλαδή προέρχονται από ηχθιοκαλλιέργειε όπου δεν περιέχουν διοξίνη. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί μπορούμε να δεχθούμε την συνέχιση της εξαίρεσης υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι απαγορεύεται η εξαγωγή. Διότι δεν μπορώ να εξάγω ένα ψάρι σε μια χώρα όπου οφείλουν να τηρούνται οι ε, περιορισμοί ναι, μεν για τη Σουηδία να μπορεί να κυκλοφορεί το ψάρι αυτό, αλλά ως εξαγωγή δεν το βλέπω. Δεν μπορεί δηλαδή να χορηγηθεί η εξαίρεση και μέσω της εξαιρέσεως μετά να μπορεί να φτάσει το προϊόν αυτό σε όλες τις ε, ε, υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί λοιπόν πρέπει να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιτρέπεται εξαγωγή. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να είναι πρόβλημα, ούτε θεωρώ ότι οι Σουηδέ και οι Σουηδοί συνάδελφοί μα αυτοδηλητηριάζονται, άλλωστε εδώ που τους βλέπω γύρω γύρω όλοι φαίνεται να χαίρουν άκρα υγεία. Ε, ευχαριστώ, θα ήθελα να απευθύνω το καλό ορίσατε σε μια ομάδα που εκπροσωπεί μη κρατικέ οργανώσεις από την Αυστρία και που ήρθαν να παρακολουθήσουν σήμερα την συνεδρίασή μα. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν προσκληθεί από την κυρία Κάριν Κάλενμπαχ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ο κύριος Κρήτον Αρσέλης. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω οι επισκέπτες μας να μην τρομάξουν από αυτά που ακούν εδώ. τα όσα προτείνει η κυρία Γουέσταν στην ουσία αποτελούν μια λογική πρόταση, δηλαδή να διατηρηθεί ένα παραδοσιακό προϊόν με ευθύνη της χώρας μέλους, αλλά δεν είναι λογικό να συνεχίσει η αλληλεία για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με αυτό το μεταποιημένο παραδοσιακό προϊόν. Ακόμα και αν, υπάρχουν, αν υπάρχει απαραίτητη ενημέρωση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Εάν δηλαδή το προϊόν μένει τελικά στην χώρα ή όχι. Δεν ε, μέμφωμαι βέβαια ότι η Σουηδία ούτε τη Φιλανδία. Το πρόβλημα θεωρώ ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόβλημα είναι διότι περνούμε από το ένα τροφιμικό σκάνδαλο στο άλλο στην Ευρώπη. Το πρόσφατο θέμα με το βακτήριο ε κόλλη στη Γερμανία ήταν ένα βαρύτατο πλήγμα στις εξαγωγές ε, προϊόντων και μιλώ για προϊόντα της εξαγωγής ε, αγροτικών προϊόντων από τις νότιες χώρες και μιλούμε για ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Πώς λοιπόν σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει περαιτέρω απώλεια αξιοπιστίας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες λόγω των αποφάσεών της. Γιατί είναι θέμα αν υπάρχει σκάνδαλο διότι δεν ελέγξαμε κάτι και είναι δύσκολο να προκύψει ένα τροφιμικό σκάνδαλο επειδή εγκρίναμε μία εξαίρεση γνωρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει συνέπειες. Εδώ βέβαια τίθεται πολλά θέματα. Εξαρτώμαστε από την κοινή αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε κάθε χώρα μέλος να εκτελεί τα καθήκοντά της ώστε προϊόντα που εγκρίνονται σε μια χώρα να είναι ασφαλή και για κατανάλωση από, από πολίτες άλλων χωρών. Και αυτή την ε, εμπιστοσύνη πρέπει να την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Ο, ο κύριος Φιέλνερ είπε κάτι για τη φέτα. Άκουσε Κρίστοφε, εγώ θα ήθελα ε, ε, εγώ δεν θα ήθελα μάλλον οι Έλληνες να τρώνε φέτα εάν αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Είναι σαφές αυτό. Και η Σουηδία τα πάει πολύ καλά. Η οικονομία που πάει πολύ καλά τώρα. Εάν δεν μπορεί τώρα να λάβει ε, μέτρα για την προστασία των πολιτών της, τότε πότε η οικονομία ε, πάει κυκλικά. Θα το κάνετε όταν η οικονομία σας τα πάει άσχημα. Έχετε, έχετε λοιπόν την ευθύνη. Έτσι λοιπόν απευθύνω ε, έκκληση πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιτρέψει άλλη εξαίρεση και πέραν των όσων είπε η κυρία Βέστλον, δηλαδή μόνο για το συγκεκριμένο παραδοσιακό προϊόν και ακόμη και γι' αυτό με επαρκής ελέγχους και ενημέρωση. Σας ευχαριστώ, η κυρία Μακάβαν, μετά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν απαντήσατε στην κυρία Westland, Westland μάλλον, είπατε ότι είδατε την έκθεση της ε, Σουηδικής ε, Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων. Αυτή τέλος πάντων η Βαλτική Ομάδα Εργασίας, η Ομάδα Εργασίας για τη Βαλτική, από ποια μέλη συναπαρτίζεται, διότι εφόσον υπάρχει έκθεση από τις αρμόδιες ειδικές αρχές, θεωρώ ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η πρώτη πηγή πληροφοριών σας. Ποια είναι αυτά τα μέλη, τέλος πάντων, της ομάδας της Βαλτικής. Και φαίνεται πως υπήρξαν αναφορές στην ε, Σουηδία σχετικά με εξαγωγές προς άλλες χώρες και ιδίως στην Γαλλία. Τα είπαν αυτά οι Γαλλίδες συνάδελφοι πριν. Τα διερεύνησε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα διερεύνησε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θέλω να μάθω διότι είπατε ότι προεξαετίας κάνατε μια έρευνα αλλά εξαετία είναι πολύ καιρό. αν κάνετε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο του χρόνου ίσως θα είναι έντονη η έλεγχη τότε μετά από τη σημερινή συζήτηση αλλά τι θα γίνει μετά από πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ως ε, σκοπό να διευκολύνει εξέβρεση διπλωματικών λύσεων όταν ε, οι Βρετανοί είχαν ε, το πρόβλημα του BSC και δεν μπορούσαν πλέον να ε, καταναλώνουν κρέας με το κόκαλο. Εγώ θυμόμαι ότι όταν ήμουν παιδί βγάζαμε το μεδούλι από τα κόκαλα και το τρώγαμε με ψωμί. Αυτά τα πράγματα απαγορεύονται πλέον τώρα. Θέλετε να απαντήσετε, να λάβετε το λόγο τώρα, κυρία Βέστλουντ μετά θα μου, το, θα μου δώσει το λόγο μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, έχω πάντω μια σύντομη ερώτηση, αν μπορούν να την απαντήσουν, να την απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Σουηδική Εύσα δεν ήθελε εξαίρεση. Η εξαίρεση φαίνεται πως δόθηκε μετά και μετά μάλιστα από διαβούλευση με την βιομηχανία. Αυτό είναι σύνηθε στην ευρωπαϊκή πολιτική για τα τρόφιμα και πώς θα ε, επηρεαστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όταν βγαίνει η ΕΦΣΑ και λέει ότι το προϊόν δεν είναι ασφαλές και ότι προκαλεί ζημιά πολλά, σε πολλά μικρά παιδιά και μωρά μέσα στην κοιλιά της μάνας τους, Αυτά συμβαίνουν, ε, είναι σύνηθες αυτό στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πριν η κυρία Κράτσα Μπίλτ θέλει ακόμα κάτι να πει. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να παρατείνουμε τη συζήτηση, αλλά δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, δεν είναι θέμα χιλιάδων παιδιών. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει, ώστε όλοι μας εδώ να ξέρουμε, τα ακριβή στοιχεία. Πόσες γυναίκες δηλαδή και πόσα παιδιά επηρεάζονται. Διότι πρέπει να μιλάμε με στοιχεία συγκεκριμένα και όχι όπως κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες ε, που τρομάζουν τον κόσμο. Δεύτερον, όλοι συμφωνούμε ότι η ενημέρωση είναι το στοιχείο κλειδί και ότι χρειάζονται σωστές ε, προτάσεις και συστάσεις από τους αρμόδιους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε να είναι αυστηρές, αυστηροί οι έλεγχοι, αυστηροί οι κανόνες, να έχουμε ε, καλές ε, συστάσεις και καλή ενημέρωση του κόσμου. Ένα πράγμα θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ η πρόταση της κυρίας δεν είναι ρεαλιστική. Γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις την ε, ξινή ρέγα από την υπόλοιπη ρέγα και το σολομό. Όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Γιατί δεν μιλάμε εδώ για τη βιομηχανία, μιλάμε για του σαλίσμα πήγατε στα, στις περιοχές εκείνες, κυρία Βέσλουντ. Είδατε ότι έχουν ένα παλιό σκάφος και ψαρεύουν εκεί. Μιλάμε για παράκτη αλεία. Δεν μιλάμε για μεγάλη κλίμακα αλεία, δεν μιλάμε για τα μεγάλα λόμπι τη αλείας. Αυτοί οι μικροί δεν θα επιβιώσουν. Αν είναι υποχρεωμένοι να αλλιεύουν μόνο ρέγγα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μεταπηθεί σε ξινή ρέγγα, δεν θα επιβιώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε. Η εξαίρεση πρέπει να είναι η πλήρηση καθόλου. Γιατί αλλιώ δεν είναι εφαρμόσιμη η πρότασή σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ωραία. Τώρα ε, οι κυρίες Χάση, και η κυρία Μπέρεντ πριν την Κομισιόν. Μα ήθελα να πάρω το λόγο, λέει η κυρία Βέσλοντ, γιατί αυτό που είπε είναι ψέμα για μένα. Και ευχαρίστω να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να πει και όχι αυτά που είπε η κυρία Κατσαμπίλτ. Η κυρία Χάση και η κυρία Μπέρεντ και μετά η Κομισιόν. Κυρία Χάση, ευχαριστώ. Τρία σημεία έχω να αναφέρω. Πρώτον, υπάρχουν παραδοσιακά πιάτα που βασίζονται στη Βαλτική Ρέγκα, στη Φιλανδία. Δεν άκουσα όμως ποτέ στη Φιλανδία κάτι που να λέει ότι χρειάζεται η μεγάλη ρέγκα της Βαλτικής για το φαγητό αυτό. Αν περιορίσουμε το μέγεθος της ρέγας που χρειαζόμαστε για ανθρώπινη κατανάλωση, θα όλο το πρόβλημα όσον αφορά τις διατροφικές παραδόσεις στη Φιλανδία με βαλτικό ψάρι. Δεύτερον, πριν από 10 χρόνια ένα από τα επιχειρήματα της Φιλανδίας ήταν όπως αυτό που ακούσαμε σήμερα από τη Σουηδία, ότι δηλαδή η... τα ποσοστά διοξίνης στους φυλαδούς είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση όταν ε, είδα τα ποσοστά διοξίνης στην Βαλτική Ρέγγα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά ήταν ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της διοξίνης δηλαδή που παίρνουμε. Η... Το αρμόδιο Υπουργείο της Φιλανδίας ε, βέβαια λέει υπέρ της παράτασης της εξαίρεσης ότι καλά-καλά δεν έχουν επιχειρήματα για τον Άγριο Σολομό. Ναι, μεν για τη Ρέγκα, αλλά όχι για τον Σολομό. Ευχαριστούμε. Ντάκμα Πέρεντ. Επανήλθε τρεις φορές η Σουηδή συναδελφός μας. Ας μιλήσω κι εγώ μια δεύτερη φορά. Ναι, λοιπόν, πράγματι, μας ενδιαφέρει η απασχόληση να διατηρείται σε δύσκολες συνθήκες και θυμούμε ότι είχαμε πρόβλημα σχετικά με την θερμοκρασία, εσωτερική θερμοκρασία των ψαριών που αλλιεύονταν για παράδειγμα στη Μεσόγειο και είχαμε πει ότι πρέπει να επιτευθεί χαμηλότερη θερμοκρασία, εσωτερική θερμοκρασία του ψαριού μία ώρα μετά την αλία τους. Αυτό θα είχε πετάξει έξω από την απασχόληση του μισού πορτογάλου ψαράδε. Αλλά απαιτήσαμε, διότι ήταν θέμα, το απαιτήσαμε διότι ήταν θέμα ασφάλεια των τροφίμων. Αυτά λοιπόν αναγκάζονται οι ψαράδε να προσαρμόζονται. Να, συνεχίσετε, να, ε, να μας λέτε τώρα ότι πρέπει να συνεχίσουμε μια πρακτική που δηλητηριάζει τον κόσμο μόνο και μόνο για να διατηρηθεί η απασχόληση. Θα έλεγα ότι είναι μια προσέγγιση ενδιαφέρουσα, αλλά δεν πιστεύω να συμφωνήσουν όλοι και ελπίζω άλλοι συνάδελφοι του Λαϊκού Κόμματος, όπω ο κ. Γκροστέτ, να φάρουν ε, τα πράγματα στην θέση του με τι παρεμβάσει του. Και ε, μια άλλη συνάδελφό μου που μου φάνηκε πιο οπορτουνίστρια. Θα ήθελα να μάθω εγώ πόσα ψάρια πιάνονται, πόσε ρέγγε ε, ψαρεύονται στην Σουηδία και Φιλανδία, άγρια και άλλα που εμπίπτουν στην εξαίρεση, διότι όταν το μάθουμε αυτό θα μάθουμε πόσα καταναλώνουν τις χώρες αυτές αφού λέτε ότι δεν εξάγονται. Αν, έχετε, αν γνωρίζετε το, τα ποσά αυτά, τότε θα γνωρίζουμε. Βέβαια, σε ορισμένες περιοχές παραθαλάσσιες οι άνθρωποι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρέγγας. Αν δεν τα έχουν τα στοιχεία αυτά οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ας μας τα πούνε κάποια στιγμή άλλη αργότερα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την συζήτηση. Θα δώσω το λόγο πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, αγαπητέ κύριε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν ε, μεγάλο ο κατάλογο των ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να απαντήσω σε όλε. Θα προσπαθήσω να τι ομαδοποιήσω. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω, γιατί θεωρώ ότι υπήρξε κάποια παρανόηση εδώ. Η τωρινή πρόταση δεν επικεντρώνεται σε εξαίρεση για την ξινή όπου υπάρχει και αναφορά στην ετικέτα της κονσέρβας. Μιλάμε και για τον άγρο σολομό και για άλλα είδη γιατί άκουσα κάποιοι βουλευτέ να ζητούν την εξαίρεση μόνο για την ξινή ρέγγα, ενώ άλλοι να λένε ότι χρειάζεται και για άλλα προϊόντα η εξαίρεση. Η ανάγκη και η αίτηση για την εξαίρεση προήλθε τα ίδια τα κράτη-μέλη, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Ζήτησαν την παράταση της ισχύουσας εξαίρεσης. Αυτό συζητήθηκε και στην ομάδα εργασίας της Βαλτικής. Και επειδή με ρωτήσατε ποιοι συμμετέχουν εδώ, συμμετέχουν κυβερνητικοί εμπειρογνώμονε. Δεν αποτελείται η ομάδα αυτή από προσώπου τη βιομηχανία, τη αλληλευτική, τη τροφική βιομηχανία. Εδώ έχουμε κυβερνητικού εμπειρογνώμονε συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τις Εθνικές Αρχές Τροφίμων. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν οι οκτώ χώρες γύρω από την Βαλτική και η προσέγγιση μας νομίζουμε ότι προσφέρει ευρεία διεξοδική εμπειρογνωμοσύνη από τις χώρες αυτές, από όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Υπήρξαν ερωτήσεις και για την ε, παρακολούθηση του όλου θέματος. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα επίπεδα διοξίνης ε, αργά μεν μειώνονται αυτό έχουν παρακολουθήσει τα στοιχεία μας. Αυτό έχουν καταγράψει μάλλον τα στοιχεία μας. Επίσης, συζητήθηκε πολύ το θέμα του ελέγχου. Να θυμίσω ότι η εξαίρεσή μας αφορά μόνο προϊόντα τα οποία γίνονται αντικείμενο εμπορίας στις εγχώριες αγορές, εσωτερικό στη Σουηδία και την Φιλανδία. Ως τώρα, δεν έχουμε καμία ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα ψάρια δεν συμμορφώνονται με τα τωρινά επιτρεπτά επίπεδα και ότι μη συμμορφούμενα ψάρια εξήχθησαν προς άλλα κράτη-μέλη. Τέθηκε ένα ερώτημα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 300 κιλά ψάρια που εξήχθησαν προς τη Γαλλία. Δεν κοινοποιήθηκε οι Γάλλοι δεν μας το είπαν. Δεν έχω καμία πληροφορία. Δεν υπήρξε κοινοποίηση από τις γαλλικές αρχές, ούτε από, Γάλλου, από Φινλανδούς ή Σουηδούς, ότι τα ψάρια αυτά ήταν εκτός ορίων. Η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν κάθε δικαίωμα να εξάγουν ψάρια αρκεί να γίνονται σεβαστά τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να απαντήσω εμέσω λοιπόν στην ερώτηση για τα 300 κιλά, δεν το παρακολουθήσαμε το θέμα διότι δεν το γνωρίζαμε. Μέχρι να τεθεί το ερώτημα της κυρίας Βέστλουν δεν είχαμε ιδέα. What uh, the commission will do, will do next. Τι θα κάνει μετά, μας ρωτήσατε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα εδώ να θυμίσω ότι επιθεωρήσεις έγιναν από το Γραφείο Τροφίμων, από την Υπηρεσία Μάλλον Τροφίμων και ιατρικών θεμάτων από το 2005. Είπα ότι εντοπίστηκαν τότε ανεπάρκειες και ελλείψεις. Όμως να ξέρουμε και ποια είναι η πρακτική αυτού του, αυτής της υπηρεσίας. Μόλις διαπιστωθούν ανεπάρκειες κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ξεκινά διάλογο, συζήτηση με την ε, ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή η υπηρεσία ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες. Οι συστάσεις που έγιναν από τους επιθεωρητές, από την, την ιατρική τέλο πάντων υπηρεσία προς τους Σουηδούς ε, ακολουθήθηκαν από τις Σουηδικές αρχές. Οπότε θα εξακολουθήσουμε, θα εξακολουθήσουμε να τονίζουμε τη σημασία της υλοποίησης των ε, αυστηρών ε, προδιαγραφών, ιδίω ως προς την ενημέρωση, αλλά αυτό είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Δική τους είναι η εξαίρεση γιατί δική τους την αγορά, αυτοί πρέπει να ενημερώσουν τους καταναλωτές τους. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση και αντίδραση σε μια παρέμβαση βουλευτού εδώ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γνωστή για το πόσο αρνείται εξαιρέσει. Δεν τις δίνουμε έτσι τις εξαιρέσει. Υπήρξαν και άλλες αιτήσει εξαίρεση από βαλτικέ χώρε που απορρίφθηκαν. Για άλλη ουσία ζητήθηκε και αύξηση των ορίων, όχι μόνο για τις ε, σκανδιναβικές χώρες, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε απαγόρευση εξαγωγή των προϊόντων αυτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό γιατί είχαμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τα άλλα 26 κράτη-μέλη. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, εδώ έχουμε απόφαση τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ε, εφαρμόζουν την εξαίρεση αυτή, διασφαλίζοντα βέβαια ότι πληρούν τι προποθέσει. Δεν έχω στοιχεία για το ποσό, τις ποσότητες αλλιευμάτων ε, στη Βαλτική θάλασσα ή για τις ποσότητες αλλιευμάτων που καλύπτει η εξαίρεση. Αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις λάβουμε είτε από τις Σουηδικές αρχές, δηλαδή τις αρχές του κράτους μέλους, ή τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Αλλά το συνολικό ποσό δεν μας δείχνει κάποιο συμπέρασμα για το τι εξαγωγές γίνονται. Μιλάμε πάντοτε για ψάρια τα οποία δεν ξεπερνούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια διοξίνης. Δεν ξέρω αν κάτι ξέχασα. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να απαντήσω έτσι κι Ευχαριστούμε. Θα, μπορούσατε, θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ακριβείς. μας λέτε οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας εάν ετήθηκαν την εξαίρεση αυτή, για ποια είδη ψαριών συγκεκριμένα τη ζήτησαν την εξαίρεση. The derogation... Η εξαίρεση αφορούσε τη βαλτική ρέγγα που ξεπερνούσε τα 17 εκατοστά, το Σολομό, την πέστροφα και άλλα δύο είδη ψαριών, για είδη βακαλα... γάδου ε, εν γέννη. Pani Magrewa na, na koniec, Pani Ένα πράγμα ξεχάσατε, Επιτροπή. Σας ρώτησα τι έγινε με την Μάλλον υπάρχει εδώ μια αναφορά στην προφορική ερώτηση για μια μελέτη από τη Σουηδική Αρχή Τροφίμων. Στην ομάδα εργασία τη συζητήσατε την μελέτη αυτή. Η κυρία Ροτμπέρεντ, με συγχωρείτε πρόεδρε. από το 2005 πότε ξαναπήγε ο ΦΑΟ στην Σουηδία και Φινλανδία. Κύριε Φιέλνερ, ούτε εγώ θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Απλώς έχω δύο αριθμούς στα χέρια μου. Για τους τόνους ψαριών που αλλιεύτηκαν βάσει της εξαίρεσης. Είναι χίλιοι τόνοι για τη ρέγγα, υπό την εξαίρεση, από του οποίους το 17-19% ε, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ξινής ρέγκας, ενώ για το Σολομό μιλάμε για 320 τόνους μόνον. Η ετήσια κατανάλωση στη Σουηδία λοιπόν είναι 13 γραμμάρια ανά, 30 μάλλον γραμμάρια ανά άτομο. Και εδώ υπόθηκε ότι η Επιτροπή δεν είχε πληροφορίες. Ότι ενημερώθηκε και από το ίδιο άρθρο που ενημερώθηκε η κυρία Βέστλουν. Μα οι σουηδικέ τοπικέ αρχέ δεν μπόρεσαν να βρουν πληροφορίε, Έκαναν έρευνα και δεν είχαν αποδείξει ότι υπήρξε αυτή η εξαγωγή. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Σα ευχαριστούμε κύριε Φιέλνερ. Κλείνουμε μάλλον τη συζήτηση για το θέμα αυτό στην παρούσα φάση. Κυρία Βέστλουντ. Θα λάβω το λόγο μετά ή, δεν έχω καταλάβει ακόμη καλά. Ή να πω, να πω τώρα κάτι. Μάλιστα, τώρα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω τώρα λοιπόν αφού μου δίνετε το λόγο. Στην πρώτη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άκουσα αλλά ίσως να μην κατανόησα καλά ότι δεν είχε λάβει την έκθεση της Αρχή ασφαλεία των τροφείων, τη σου ειδική ασφαλεια των Τροφίμων, της Σουηδικής ασφαλεια των Τροφίμων, που έλεγε ότι λίγες μόνο οι οικογενειε στη Σουηδία που έχουν παιδιά είναι ενήμερες και αναγνωρίζουν το προϊόν το οποίο περιέχει διοξίνη. Στην ουσία έχω την αίσθηση ότι η Σουηδική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρύψει την ε, υπόθεση. Λέει η, Σουηδική, λέει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει λάβει την έκθεση. Εγώ όμω έστειλα η ίδια στην αρμόδια επίτροπο την έκθεση, καθώ επίση και ένα άρθρο με έναν ε, που μιλεί ένα εξαγωγέα, ένα άρθρο εφημερίδα, που λέει ότι έχει κάνει εξαγωγέ του ψαριού αυτού στην Γαλλία. Το έστειλα το άρθρο αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακούω τώρα ότι δεν την έχουν λάβει την ε, πληροφορία αυτή. Δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί η κατανάλωση με ξεκάθαρο τρόπο. Οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε ωστόσο δείχνουν ότι χιλιάδες μικρά παιδιά αλλά και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία κινδυνεύουν να καταναλώσουν υπερβολικές ποσότητες διοξίνης μέσα των ψαριών. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή, δεν υπάρχει έλεγχο. Όταν ρωτήθηκε ο αρμόδιος υπουργό ποιος φέρει την ευθύνη για την ε, παρακολούθηση της επιβολής της απαγόρευσης, δεν πήραμε απάντηση. Επίσης, όταν απευθυνθήκαμε στις τοπικές αρχές και ρωτήσαμε ποιος είναι υπεύθυνο για την ε, παρακολούθηση της απαγόρευσης, λάβαμε δεν λάβαμε απάντηση. Τώρα μαθαίνουμε ότι κάθε τοπική αρχή η οποία έχει μια ήχθη είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της απαγόρευσης εξαγωγής. Πολλά γεγονότα βεβαίως, πολλά facts πρέπει να εξεταστούν. Ουδής ισχυρίζεται ότι η διοξίνη στα ψάρια είναι πρόβλημα για όλους τους Σουηδούς. Για παράδειγμα, Σουηδοί άνδρες, ενήλικοι άνδρες δηλαδή, μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα από τα ψάρια αυτά χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, νέες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία ή έμβρια ή μικρά παιδιά, μωρά, μπορεί να υποστούν πολύ μεγάλη ζημιά. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξετάζεται το επίπεδο της διοξίνης και στο γάλα θυλασμού. Μιλούμε για αυτές τις χιλιάδες παιδιά και γυναίκες που λένε ότι καταναλώνουν πολύ βαλτική ρέγγα. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Δεν είναι βέβαια το πρόβλημα για τα πρόσωπα εκείνα που δεν τρώνε τα ψάρια αυτά, αλλά για τα πρόσωπα που τρώνε τα ψάρια αυτά και που δεν έχουν σχετική ενημέρωση και που κινδυνεύουν από σημαντικέ βαριέ επιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον επίση ότι απέναντί μα βρίσκεται μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν παρακολουθεί τα γεγονότα, τη στέλνει μάλιστα την ενημέρωση και δεν την λαμβάνει ή δεν την βρίσκει, ενώ έχουμε τη Σουηδική Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων που λέει ότι είναι κίνδυνος για το κοινό, έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μανάδες οι οποίες τρώνε τα ψάρια αυτά και παρόλα αυτά το μόνο που φαίνεται να ενδιαφέρει εδώ είναι ότι θα θυγεί ο κλάδος. Ναι, και για την ξινή ρέγγα. Εγώ δεν θέλω να σταματήσουν οι Σουηδοί να τρώνε την ξινή ρέγγα, αλλά ίδια η βιομηχανία λέει ότι δεν μπορεί να παραγάγει την ρέγγα παρά μόνο εάν αλλιεύσει ψάρια που έχουν υψηλό επίπεδο διοξίνης λόγω λίπους. Η ξινή ρέγγα, μας λένε όμως άλλοι, μπορεί να παράγεται ακόμα και με την, ε, και με την ε, άρση της εξαίρεσης. Θα είναι ίσως λίγο πιο ακριβή τότε η ξινή ρέγγα, αλλά νομίζω ότι δεν θα αποτρέψει αυτό όσους ενδιαφέρονται να την καταναλώσουν. Είναι δύσκολο βέβαια να επηρεαστεί η απόφαση αυτή, διότι η απόφαση για την εξαίρεση λαμβάνεται από ειδική επιτροπή. Πάντως ας γνωρίζουν τα μέλη της ότι όλοι τους παρακολουθούν και η Σουηδική κυβέρνηση και αυτή οφείλει να αντιδράσει και να φροντίσει να προστατεύσει τα παιδιά που κινδυνεύουν από την διοξίνη. Νομίζω το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί με κατάλληλο τρόπο στο παρελθόν σε, ένα, σε συνεντεύξεις τύπου κτλ. Διότι όλοι το περιορίζουν μονάχα στο θέμα της ξενής ρέγκας. Ενώ δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Άρα πρέπει να βελτιωθεί η ενημέρωση ώστε να κινδυνεύουν λιγότερα παιδιά. Εγώ θα επιμείνω, δεν πρόκειται να αφήσω το θέμα αυτό, να εγκαταλείψω το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να αμφισβητούνται τα στοιχεία αυτά πρέπει να φροντίσουμε ώστε η ενημέρωση να φτάνει στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται. Και ελπίζω στο μέλλον να προκύψει κάποια αλλαγή και τα πράγματα αυτά να λαμβάνονται σοβαρότερα υπόψη, γιατί μιλάμε εν τέλει για το μέλλον των παιδιών μας. Θέλω να ρωτήσω μονάχα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν να ζητήσει από τη Σουηδική Κυβέρνηση να βρει τις προφορίες. τον μαθαίνω εγώ ότι 300 κιλά από τα ψάρια αυτά εξήχθησαν στην Γαλλία προφανώς χωρίς ε, την απαραίτητη έγκριση και ότι καμία πληροφορία δεν περιλαμβάνεται για την περιεκτικότητα των ψαριών αυτών, εγώ θέλω να μάθω αν νομίζω ότι η διοξίνη αναφέρεται ως PPSD ή κάτι τέτοιο εγώ θα θέλω να, να γράφει επάνω διοξίνη. Ε, εφόσον η φιλανδική και η παράδοση επιτρέπει την κατανάλωση ψαριών που περιέχουν διοξίνη, ε, εντάξει, δική τους υπόθεση είναι, δική τους παράδοση είναι. Ως Γαλλίδα όμως θέλω οι συμπολίτε μου να είναι ενήμεροι για το τι τρώνε. Είναι δυνατόν αυτό ναι ή όχι ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φλου. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις ε, <clears throat> υπήρχαν και για σας, γι' αυτό σας δίνω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ για την έκθεση που ρωτήσατε. Εμείς δεν πήραμε την έκθεση της Σουηδικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων. Για την τελευταία ερώτηση, αν σας κατάλαβα καλά, και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει απαγόρευση εξαγωγής ηχθείων από την Σουηδία ή την Φιλανδία προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, υπάρχει θέμα άδειας ε, και λοιπά για τέτοιες εξαγωγές. Επιτρέπονται. Αλλά οι χώρες που εξάγουν και κυρίως οι χώρες που εισάγουν πρέπει να επικεντρώνονται σε ελέγχους κάθε φορά που πρόκειται για προϊόντα που έρχονται από την Σουηδία και τη Φιλανδία εφόσον το επιθυμούν. Είναι ευθύνη δηλαδή των χωρών μελών να επικεντρωθούν ή να έχουν ως προτεραιότητα του ελέγχου στα προϊόντα που θεωρούν ότι θέλουν να ελέγξουν. Και τη ΦΑΟ επίσης είπατε ότι πάει καιρός που δεν έχει πάει σε αυτές τις χώρες. Πράγματι, το 2005 είχε πάει. Το αποτέλεσμα όμως της αποστολής αυτής, παρά κάποια πράγματα που είχαν εντοπίσει, δεν είχαν ε, καταλήξει σε προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρξει νέος γύρος επισκέψεων σε αυτές τις χώρες εν ώψη νέας εξαίρεσης. Όσον αφορά τώρα τις απαιτήσει για τις ετικέτες, από όσο ξέρω, είναι θέμα προέλευσης. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα δεν βλέπω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που θέτεται πέρα από την ενημέρωση των καταναλωτών για το ότι μπορεί να περιλαμβάνουν τα προϊόντα αυτά διοξίνες ή BCB. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λίγη η συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό και ευχαριστώ πολύ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους τους συμμετέχοντες. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο αριθμός 7 στην ημερήσια διάταξη. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Περιβάλλον. Κυρίε και κύριοι, έχουμε έξι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε εδώ. Είναι ερωτήσεις μας ε, και περιμένουμε ε, απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 10 λεπτά για την κάθε ερώτηση, γιατί έχουμε μια ώρα στη διάθεσή μας και αφού είναι 6 ερωτήσεις, 10 λεπτά η καθεμία για να τελειώσουμε έγκαιρα, στις 12.30 δηλαδή πρέπει να τελειώσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ξεκινάμε λοιπόν με την ερώτηση αριθμός 1 που θέτει ο κύριος Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Πρόκειται για το REACH, Έχετε τις διάφορες πληροφορίες στους φακέλους σας. Έχουμε εδώ πέρα δύο εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάρφιν και Κάνσελ, Οπότε παρακαλώ να μας απαντήσετε. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Επειδή μου δίνετε λίγο χρόνο, θα συνοψίσω λιγάκι τις τρεις υποερωτήσεις που αναφέρονται εδώ και δεν θα μπω στις λεπτομέρειες παρόλο που είχα ετοιμάσει και πολλές λεπτομέρειες να σας μεταφέρω. Αν χρειαστεί όμως και εφόσον θέλετε θα σας προσφέρω και συμπληρωματικές απαντήσεις όποτε εσείς το επιθυμείτε. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν έχει να κάνει με ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά το REACH. Ίσως θα έπρεπε να πω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών έχει, μας έχει ενημερώσει και έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία από αυτού. Δεν θα σας αναφέρω πολλά τώρα νούμερα, θα επικεντρωθώ κυρίως στην άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά το ρίτ σε γενικές γραμμές. Το κύριο κομμάτι του REACH έχει να κάνει με δραστηριότητες της βιομηχανίας προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις ε, υποχρώσεις τους καταχώρησης. Η ε, δημιουργία, η συλλογή πληροφοριών προκειμένου να μπορούν οι διάφορες ε, επιχειρήσεις της βιομηχανίας να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να βρουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης. Μόλις συμπληρώθηκε η πρώτη, μάλλον μόλις πέρασε η πρώτη προθεσμία καταχώρησης. Πάνω ή μάλλον περίπου 25.000 υποθέσεις πήγανε στην υπηρεσία χημικών για όλες τις χημικές ουσίες για τις οποίες υπήρχε τέτοια απέτηση όσον αφορά την πρώτη προθεσμία καταχώρησης. Πρόκειται για χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες πάνω από χίλιους τόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόκειται και για διάφορες άλλες ουσίες επικίνδυνες, ε, καρκινογενείς κλπ. Στην καταχώρηση λοιπόν όλων αυτών των χημικών ουσιών έχουμε πρώτα απ' όλα τον όγκο. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου κατοχωρείται λοιπόν σήμερα. Έπειτα οι δραστηριότητες όσον αφορά αυτές τις ουσίες έχουν εντοπιστεί και έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε μέτρα διαχείρισης κινδύνου για τη, να ελέγξουμε τις ουσίες αυτές και για να ε, μπορούμε να ενημερώνουμε τους παρετέρω χρήστες ή τελικούς καταναλωτές όσον αφορά ε, τους κινδύνους αυτούς. Αναπόφευκτα αυτό οδηγεί σε μια πιο ασφαλή χρήση χημικών ουσιών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, όπως επίσης και σε ένα ε, καλύτερο και πιο καθαρό περιβάλλον. Είμαστε όμως στην αρχή της διαδικασίας, γιατί η καταχώρηση δεν είναι παρά το σημείο εκκίνησης όσον αφορά τα χημικά τα οποία μπαίνουν μέσα στο σύστημα του REACH. Στη συνέχεια έχουμε άλλες δύο σημαντικές προθεσμίες καταχώρησης που είναι το 2013 για πάνω από 100 τόνους και το 2018 για χημικές ουσίες ανάμεσα στον έναν και στους 100 τόνους. Η διαδικασία αξιολόγησης τώρα ε, προχωράει. Βελτιώνεται και επιταχύνεται. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών έχει ένα χρόνο στη διάθεσή της για να φέρει σε πέρα τις περισσότερες δραστηριότητες αξιολόγησής της. Αυτό όμως σημαίνει ότι δουλεύουν σκληρά και ότι τα αποτελέσματα που έχουμε είναι τα αποτελέσματα των υποθέσεων που ε, άρχισαν να εξετάσουν πριν από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε λιγότερα αποτελέσματα από όσα θα έχουμε όταν ε, προχωρήσει σε κανονικό ρυθμό. Βλέπουμε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ότι το 2010 για παράδειγμα εξέτασε 273 ε, υποθέσεις καταχώρησης. Έγινε η καταχώρηση πριν από την προθεσμία όμως του Νοεμβρίου του 2010 και τότε τους τελευταίους μήνες ήταν που είχαμε τις περισσότερες καταχωρήσεις. Όσον αφορά τις άδειε. Το Φεβρουάριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε απόφαση για να προσθέσει άλλα δύο έξι χημικά μεγάλων συγκεντρώσεων από τον κατάλογο υποψήφιων προϊόντων προς άδεια. Και η Επιτροπή είναι στη διαδικασία εξέτασης και παρακολουθεί την διαδικασία έτσι όπως προβλέπεται μέσω των ρυθμιστικών επιτροπών για άλλε 8 ουσίες από τον κατάλογο αυτό προϊόντο που θα μπορούσαν να προσθεθούν στις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προς αδειοδότηση. Συνολικά πρόκειται για 46 ουσίες και η Επιτροπή την προηγούμενη χρονιά ότι υπάρχουν και άλλες 90 ουσίες που θα έπρεπε να προσθεθούν στον κατάλογο με υποψήφιες ουσίες μέχρι το 2012 και τέλος θέλουμε σαν τελικό στόχο να συμπεριλάβουμε όλες τις ουσίες υψηλής περιεκτικότητας μέχρι το 2020. Προς το παρόν και πριν από 21 μέρες έληξε η προθεσμία για τις πρώτες κοινοποίησεις για ουσίες ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης και άρχισε να ισχύει υποχρέωση για την βιομηχανία, τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς των προϊόντων αυτών να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών εφόσον υπάρχει ένα προϊόν το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 0,1% επικίνδυνης ε, ουσίας. Κατά συνέπεια, έξι μήνες μετά από κάθε νέα ουσία που προστίθεται στον κατάλογο, η υποχρέωση αυτή αρχίζει να ισχύει για τη συγκεκριμένη ουσία. Για τους περιορισμούς τώρα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τελικό σώμα που κάνει προτάσεις για περιορισμό ουσιών. Μετά από πολλή δουλειά βέβαια. Έχουμε περιορίσει πολλές ουσίες πρόσφατα. Για το κάδμιο, για ό,τι περιλαμβάνει κάδμιο η εφαρμογή προσφεύγει σε ένα καινούριο σώμα, το Φόρουμ όπως ονομάζεται, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και έχει προχωρήσει στις πρώτες συντονιστικές δραστηριότητες υποχρέωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντοπίζουμε λοιπόν τα διάφορα προβλήματα, τα αναφέρουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, συμμετέχουν και καλύπτονται από τις απαιτήσει καταχώρησης έχουν μια προθεσμία για καταχώρηση που είναι το 2018. Όσο χαμηλότερο όγκο χημικών, τόσο περισσότερο θεωρούμε ότι θα συμμετέχουν αργότερα περισσότερες επιχειρήσεις. Είπαμε ότι είχαμε και πέρυσι μια προθεσμία που έληξε και το 2013 άλλη μία. Πιστεύουμε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν θα είναι μικρότερο από αυτό που θα έχουμε το 2018. Έτσι λοιπόν αρχικά φτιάξαμε μια ομάδα επαφής για να προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταχώρησης, πρώτα απ' όλα την περσινή. Η ομάδα αυτή θα συνεχίσει τη δουλειά της μέχρι τη λήξη της επόμενης προθεσμίας και ένα από τα καθήκοντά της είναι να συλλέγει πληροφορίες, ιδιαίτερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα προβλήματα στην πράξη που αντιμετωπίζουν προκειμένου να ετοιμάσουν τους φακέλους που υποβάλλουν για καταχώρηση. Αυτή η ομάδα επαφής εξετάζει λοιπόν τα πρακτικά προβλήματα και προσπαθεί να βρίσκει πάντα ε, πρακτικές, καλές και ικανοποιητικές λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, όσον αφορά την αναθεώρηση του REACH, εδώ θα είμαι σύντομος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία ιστοσελίδα Εκεί ενημερώνουμε για την πρόοδο που επιτυχάνεται όσον αφορά την αναθεώρηση του REACH. Η ιδιαίτερη αναθεώρηση αυτή έχει να κάνει με τα τρία στοιχεία που απαιτεί το REACH, που είναι αναθεώρηση της υπηρεσίας χημικών, των απαιτήσεων πληροφόρησης από έναν μέχρι 10 τόνους χημικά και αναθεώρηση βέβαια του εύρους της νομοθεσίας και να δούμε τι επικαλύπτεται από άλλη νομοθεσία. Επιπλέον πάντως προχωράμε και σε διάφορες μελέτες για να δούμε τι επιπτώσεις έχει το Ρίτ στην ανταγωνιστικότητα, στο κόστος, στην καινοτομία αλλά και τα ωφέλη για την υγεία από το Ρίτ. Εξετάζουμε επίσης διάφορες παράλληλες ανεξάρτητες μελέτες μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξίζει τον κόπο επίσης να πούμε ότι ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα διαβουλεύσεων με ε, διασκέψεις όσον αφορά την αναθεώρηση για του χρόνου. Τελειώνοντας την έκθεση τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς. Τέλος, τα καυτά νέα της ημέρας είναι ότι σήμερα προσθέθηκαν άλλες 7 ουσίες στον κατάλογο με τις ε, ενδεχομένως επικίνδυνες ε, ουσίες. Σας τα είπα περιληπτικά και ελπίζω να αρκούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Φλόρενς. Μία σύντομη ερώτηση. Θυμούμε όταν συζητούσαμε την οδηγία REACH συμμετείχαν ορισμένοι συνάδελφοι που έλεγαν ότι η καταχώρηση αναφέρονταν σε 15-20 χιλιάδες προϊόντα, τώρα μιλείτε για 25 γνωρίζετε από πού προέρχονται ή ήταν οι πληροφορίες εκείνες τότε εσφαλμένες. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, είχαμε πει τότε ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα απαλλαγούν βαρών με την έννοια ότι θα πούμε ότι ένα συστατικό σημαίνει μια έγκριση. Εάν λοιπόν 100 ε, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο συστατικό, μια ουσία, θα χρειάζονται μία έγκριση. Ε, αυτό ισχύει ή όχι. Ευχαριστώ για την ε, ιδιαίτερα περιεκτική σας ε, έκθεση. Μιλήσατε για 136, λέει ο κ. Σλάιτερ, για πριν από δύο χρόνια τώρα. Έχετε φτάσει στις 53. Για τα ενδιάμεσα, 86% των ουσιών ήταν στο καθεστώς αυτό των ενδιάμεσων. Επίσης 64% των φακέλων, των ντοσιέ που εξετάστηκαν ήταν ελληματικά. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο αριθμό ντοσιέ που θα περάσουν θα, κάπως λαθρέα. Θα μπουν δηλαδή το εφόσον έχετε ένα κατόφλι 5%. Δεν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα τώρα. Δεν είναι σωστό να μάθουν οι επιχειρήσεις από την αρχή να συνθέτουν του φακέλους, τα δοσία σωστά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουμε και το πρόβλημα των ψευδών μικρομεσών επιχειρήσεων. Με ποια στατική θα το αντιμετωπίσετε. Χρειαζόμαστε επίση έλεγχο περισσότερων φακέλων. ...20% αποδίδει σήμερα, ενώ το σχέδιο προβόταν 28% του προσωπικού επιτόπου. Εσείς κύριε Χάνσιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις πρόσθετες ερωτήσεις σας που ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω ικανοποιητικά. Και θα αρχίσω με το θέμα των αριθμών του κύριου Φλόρενς. ήταν σχεδόν 25.000 ντοσχέ καταχώρησης που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που παράγει μια ουσία που εμπίπτει στα κριτήρια καταχώρησης μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να υποβάλει ντοσχέ καταχώρησης και κατά μέσον όρο 7 έως 8 δοσία καταχώρησης ανά ουσία. Αυτές οι 25.000 λοιπόν αναφέρονται σε περίπου 3.000 ουσίες συστατικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις εκτιμήσεις μας στο χρονικό αυτό σημείο, οι εκτιμήσεις που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ΡΙΤΣ και τις αναθεώρησε το 2005 νομίζω, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Δελτίου, ήταν ε, νομίζω αρκετά σωστές. Τώρα εργαζόμαστε για, επί των ουσιών εκείνων που γνωρίζαμε καλύτερα. Μεγαλύτερες αβεβαιότητες είχαμε για την επόμενη προθεσμία καταχώρησης. Πώς λειτουργεί τώρα το μία καταχώρηση, μία ουσία και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η καταχώρηση λειτουργήσε ήταν και μια ένδειξη ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν. Η Directors Contact Group εργάστηκε σκληρά με τον κλάδο και ο κλάδος εργάστηκε σκληρά για τις καταχωρήσεις και για να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε συνεργασία μαζί τους. Δεν θέλω λοιπόν να μειώσω την αξία των προσπαθειών που κατέβαλε ο κλάδος και για την συνεργασία και για την διατήρηση επαφών μια πρωτοφανής συνεργασία στην Ευρώπη και ιδίω για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Λάβαμε λοιπόν τις ε, καταχωρήσεις, λειτουργήσε το σύστημα και αυτό δείχνει ότι τα προβλήματα δεν ήταν αξεπέραστα. Θα ασχοληθούμε σοβαρά να αναλύσουμε σε συνεργασία με την βιομηχανία τα προβλήματα και να εξομαλύνουμε βεβαίως όσο γίνεται περισσότερο μέχρι την επόμενη ε, προθεσμία και μάλιστα την τελευταία όπου αναμένεται ακόμα περισσότερε μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να συμμετάσχουν. Τα τελευταία τέσσερα θέματα στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του 2012 για ορισμένες ουσίες εργαζόμαστε επ' αυτής, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει αναγνωρίζουμε επίσης ότι οι χώρες μέλη έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην πρόταση ουσιών για να μπουν στη λίστα των υποψηφίων και συνεργαζόμαστε και με τις χώρες μέλη αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα επιτύχουμε τον στόχο αυτό που έχουμε αναλάβει να επιτύχουμε. Το 68% των ενδιαμέσων που ανακοίνωσε η ΕΚΑ στην ιστοσελίδα της που πιθανώς να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσει για να αναγνωριστούν ως ενδιάμεσες. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την ΕΚΑ τώρα για να κατανοήσουμε σε ποια βάση βασίζονται αυτές οι ενδείξεις. Η ΕΚΑ ίδια λέει στην ιστοσελίδα της ότι πρόκειται για ένα προκαταρκτικό πόρισμα, αλλά στον χώρο αυτό συνεργαζόμαστε ενεργά για να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα και για να χαρτογραφήσουμε τους καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Ε, υπάρχει, μια, ε, υπάρχει ένας αριθμός ε, τρόπων αντιμετώπισης βεβαίως και επιβολής αλλά και άλλων. Πάντως το πρόβλημα αυτό μας απασχολεί και βεβαίως ναι, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το 64% των ελληματικών ντοσιέ, το ίδιο εδώ πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα ακριβώς η μάλλον πρέπει να κατανοήσει αλλά και εμείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πού ακριβώς ε, ε, εντοπίζονται οι ελλείψεις και με ποια στατική θα τις αντιμετωπίσουμε. Το 5% βέβαια αποτελεί μια επιλογή που μας έδωσε ο νομοθέτης για να το εξετάσουμε, να εξετάσουμε δηλαδή τα ελληματικά ντοσίε. Αλλά πρώτα μας χρειάζεται μια στέρεα βάση για να το κάνουμε αυτό. Και τέλος ό,τι αφορά τις ψεύδο μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ΕΚΑ κάνει πολλή δουλειά γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της διότι ε, τα τέλη είναι περιορισμένα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΚΑ λοιπόν έχει ενδιαφέρον να κάνει μια σε βάθος ανάλυση για να εντοπίσει τις ψευδείς αυτές μιμιέ και η ΕΚΑ το κάνει αυτό και άλλοι, και άλλοι παράγοντες βέβαια αλλά γνωρίζουμε και εμεί τη ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ΕΚΑ ε, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πολύ μεστή απάντηση και ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Το πρώτο μας πήρε 20 λεπτά. Ίσως μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένες, πιο σύντομες απαντήσεις στο επόμενο. Ερώτηση δηλαδή του κυρίου Βιτόριο Πρόντι και την απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στο ερώτημα, να σας δώσω κάποια στοιχεία για το πώς έχει εξελιχθεί ως τώρα η νομοθεσία. Και εξηγώντας το πώς έχει η νομοθεσία θα σας απαντήσω και στο ερώτημα το πρόγραμμα αναθεώρησης για τα διεκτώνα καλύπτεται από τον κανονισμό της Επιτροπής 1451 το 2007. Υπάρχουν τρεις, 300 ουσίες που καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό και με το πρόγραμμα αναθεώρησης τι συμβαίνει. Οι εταιρείε που βάλουν ένα λεπτομερές αυτό το τα κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει για κάθε ουσία να εντοπίζουν και να καταγράφουν είναι ουσιαστικά οι αρχές ε, αδειοδότησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Αυτές εξετάζουν λοιπόν τα ντοσιά και τέλος υποβάλλουν και την ε, έκθεση, την ε, τοποθέτησή τους δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της αποτίμησης της, του ντοσιέ. Έπειτα έχουμε περαιτέρω συζητήσει με το κάτω μέλο και γίνεται, λαμβάνεται η απόφαση αν θα περιληφθεί στον γενικότερο κατάλογο των ουσιών η εν λόγω ουσία ή όχι. Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αναθεώρηση, είδαμε ότι στο 90% των περιπτώσεων μία μόνο εταιρεία, υπέβαλε, ένας μονοφορέας υπέβαλε κάθε φορά ένα ντοσιέ. Ε, ήταν όμιλος ή ήταν μία και μόνο εταιρεία. Ε, ήταν λοιπόν κάθε φορά ένα αυτό που έβαλε τον Τοσιά, έτσι καθοριζόταν και το κόστο. Τώρα, όταν ήταν πάνω από μία οντότητα, ε, εδώ ο κανονισμό προβλέπει ότι πρέπει να γίνει εύλογη προσπάθεια συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων εταιριών, δύο, τριών, όσοι είναι, για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Σύμφωνα με τα δικά μα τα αρχεία, μόνον πέντε ουσίες τι οποίε εμεί γνωρίζουμε, αντιμετώπισαν δυσκολίε στην ανταλλαγή δεδομένων. Οι πέντε αυτές ουσίες, οι πέντε αυτές υποθέσεις αφορούσαν τις ίδιε ακριβώ ε, ακριβώς δύο εταιρείε. Η μία είναι μία μεταπητική εταιρεία εντός Ένωση και η άλλη εκτός. Ε, υπάρχουν κοινοποίησει και για τι πέντε περιπτώσει. Στην πρώτη περίπτωση επιτέχθη συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη δεύτερη περίπτωση η αρμόδια αρχή, η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή, θεώρησε ότι όλε οι εύλογε προσπάθειε για την ανταλλαγή δεδομένων έγιναν και από τι δύο πλευρέ, όμω εδώ δεν συμφώνησαν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου βρισκόταν η Ευρωπαϊκή Μεταποιητική Εταιρεία. Ε, έτσι λοιπόν υποβλήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης αξιολόγηση της αμμόδιας αρχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά τα της προσφυγής αυτής. Ακόμη έχουμε συζητήσεις με την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξέταση των τοσχέ αυτή και για το πόσο δεν επετέφθη συμφωνία ανταλλαγή δεδομένων. Για τι άλλε υποθέσει, οι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε είναι ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίε για την επίτευξη συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων και ακόμη δεν έχουμε λάβει στοιχεία για κάποιο περαιτέρω βήμα. Για τις 300 λοιπόν ουσίες του προγράμματος αναθεώρησης εντοπίστηκαν μόνο 5 που υπήρχαν δυσκολίες για την ανταλλαγή δεδομένων και μία όπου τελικά επετεύχθη η συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων. Τέσσερι στην ουσία λοιπόν, αυτέ που αντιμετωπίζουν δυσκολίε και αυτέ αφορούν και σε όλε τι περιπτώσει τι ίδιε δύο εταιρείε. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τις εν λόγω ουσίες και τις εταιρείε. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προς συνέπειες, διότι ο κανονισμός για τα βιοκτώνα ορίζει ότι ακόμη και εταιρείε που έχουν διαφορά ω προ την ανταλλαγή των δεδομένων μπορούν να συνεχίζουν να εμπορεύονται προϊόντα με τι ενεργές αυτέ ουσίε τουλάχιστον για δύο χρόνια μετά τη συμπερίληψη των εν λόγω ουσιών στο γενικότερο κατάλογο ουσιών του παράδειγματος 1 του κανονισμού. Αυτό σημαίνει ότι στην παρούσα περίπτωση και οι πέντε αυτές ουσίες που σας ανέφερα θα συμπεριληφθούν τελικά στο παράδειγμα 1, τον κατάλογο του παράδειγματος 1 του κανονισμού, όμως τα προϊόντα των δύο εταιριών βρίσκονται ακόμη στην εμπορία γιατί για την ώρα δεν υπάρχουν πρακτικές συνέπειες εκτός από ούτε θέματα πρόσβασης των προϊόντων στην αγορά. Το πρόβλημα θα προκύψει όταν οι ουσίες θα συμπεριληφθούν έπειτα στο παράρτημα. Το νωρίτερο που θα συμβεί αυτό είναι τα μέσα του 2012 οποιαδήποτε από αυτές τις πέντε ουσίες. Άρα μέχρι το 2014 οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να έχουν υποβάλει ντοσχέ για τα προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ενεργές ουσίες. Όταν θα υποβάλουν τα ντοσχέ αυτές μπορούν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να ανταλλάξουν δεδομένα. Εάν δεν το καταφέρουν τότε μπορεί η δεύτερη εταιρεία που δεν έχει τα δεδομένα, της λείπουν τα δεδομένα, είτε να βγει εκτός αγοράς, είτε να κάνει τις υπολοιπόμενες ε, δοκιμές. Όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η νέα πρόταση κανονισμού τα βιοκτώνα που θα τη δει το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση από το Σεπτέμβριο συμπεριλαμβάνει μέτρα που υπερβαίνουν τα όσα προβλέπει η ισχύουσα οδηγία και επιτρέπει στις εταιρείε επιβάλλει μάλλον στις εταιρείε να ανταλλάσσουν μεταξύ του τα δεδομένα. Ο τωρινό κανονισμό λέει ότι μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα. Τώρα θα υποχρεώνονται με τον νέο κανονισμό. Ε, προγραμματίζουμε λοιπόν με τον νέο κανονισμό να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ ω τα μέσα του 2012 και να υλοποιείται το αργότερο από τα μέσα του 2013. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ε, οι υποχρεώσει των εταιριών για ανταλλαγή δεδομένων θα ισχύουν. Άρα οι πέντε ουσίες για τις οποίες υπάρχουν διαφορές θα καλύπτονται από τον, ε, τους κανόνες του νέου κανονισμού. Δηλαδή ό,τι προβλήματα υπάρχουν θα πρέπει ως τότε να λυθούν. Νομίζουμε λοιπόν ότι οι πέντε αυτέ εν λόγω ουσίε δεν θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα στι συγκεκριμένε εταιρείε ώστε να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Πρόντι, ευχαριστώ την Επιτροπή για τα στοιχεία που μας έδωσε. Νομίζω και έχοντας υπόψη τις διαστάσεις των εταιριών αυτή μπορεί να είναι και μια είδους εγγύηση, διασφάλιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν, διότι η κατάσταση που μας περιγράφει η Επιτροπή είναι καθυσχαστική. Θα δούμε πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν και στην πράξη. Ευχαριστώ πάντως για τις τόσες λεπτομέρειες και για την θετική προοπτική που μας δώσατε. Συνολικά θα καλυφθούν τουλάχιστον οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση για τα απόβλητα. Καλ Χάιντς Φλόρενς. Komisji głos zabierze pan Peter Ο κύριος Βέστμαν εκ μέρους της Επιτροπής. Πρόεδρε, για τον ανυπομείνοντα χρόνο και με τις αναπομείνασες ερωτήσεις θα ήθελα να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Η υλοποίηση τη νομοθεσία για τα απόβλητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια ασχοληθήκαμε με τα πολυάριθμα κενά κατά την υλοποίηση και την επιβολή του κεκτημένου αυτού. Ένα παράδειγμα είναι η απουσία υποδομών επεξεργασία των αποβλήτων σε κάποια κράτη-μέλη και ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαδεδομένη ε, χρήση παράνομων και κακοδιαχειριζόμενων χωματερών. Αυτό έχει να κάνει και μετά όσο ορίζει οδηγία πλαίσιο και μας απασχολεί μεγάλος αριθμός ε, παράνομων αποστολών αποβλήτων το 20% του συνόλου των μεταφορών που αφορούν απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το 20% παράνομες. Και αυτό έχει να κάνει και με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταφορά αποβλήτων, τι αποστολέ ε, αποβλήτων. Για να παροτρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερη συμμόρφωση με τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, έχουμε προβλέψει διάφορε δράσει. Θα τι συνοψίσω σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα ε, οργάνωσε εκδηλώσει ευαισθητοποίηση του κοινού και ενημέρωση σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να ενισχύσει την υλοποίηση και επιβολή τη νομοθεσία για τα απόβλητα. Τα στοιχεία αυτά θέλουν να ενισχύσουν την πραγματική συνεργασία και την μεταφορά πληροφοριών για την υλοποίηση, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών άμεσα μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων. Τα στοιχεία αυτά έχουν καλύψει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποστολές αποβλήτων, τα απόβλητα και τις χωματερές. Το 2009 έως 2011, 60 ε, εκδηλώσεις αυτού του τύπου οργανώθηκαν στα κάτι μέλη. Τώρα ε, συνεχίζουμε με τον προγραμματισμό άλλων 15 εκδηλώσεων που αφορούν συγκεκριμένα τη νέα οδηγία πλαίσια για τα απόβλητα. Οδηγία που θα ολοκληρωθεί φέτος. Εδώ ε, θα προβλέπονται υποχρεώσεις για προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων και πρόληψης ε, της παραγωγής αποβλήτων. Εδώ συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε κατευθυντήριε γραμμέ για να στηρίξουμε τι εθνικέ αρμόδιε αρχέ, του οικονομικού φορεί και του ενδιαφερομένου του τομέα, ώστε να υλοποιούν καλύτερα την οδηγία περί αποβλήτων. Έχουμε διάφορε κατευθυντήριε γραμμέ, σημαντικέ κατευθυντήριε γραμμέ, ε, δημοσιευμένε στον τόπο μα, δηλαδή πώ να καταρτίζει κανεί προγράμματα διαχείριση των αποβλήτων, πώ να ανοιχνεύει και να προλαμβάνει παράνομε μεταφορέ αποβλήτων και πώ τα ουσιαστικά σημεία τη οδηγία περί αποβλήτων να τις ε, εφαρμόζει σωστά όπω την οδηγία για, το τέλος, για τα οχήματα που βρίσκονται στο τέλο τη ζωή του, για τι μπαταρίε και το καθεξή. Επίση, έχουμε δημιουργήσει ένα help desk, μια γραμμή επικοινωνία για να διευκρινίζονται οι απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα απόβλητα και αυτή η γάμπη επικοινωνία, αυτό το ε, help desk έχει ασχοληθεί με κάποια ζητήματα προτεραιότητα. Έχουμε δημοσιεύσει μάλιστα εγχειρίδιο σε σχέση με τα ζητήματα που συχνότερα ανακύπτουν στον τοπό μα. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί ε, επικεντρωνόμενο ε, στα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τα απόβλητα, καθώ και την καλύτερη και γρηγορότερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μια ηλεκτρονική πλατφόρμας που θα διατεθεί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Europa. Ε, παρά τις δράσεις αυτές όμως που ανέφερα, είναι πολλά αυτά που απομένει να γίνουν. Χρειάζονται περισσότερες δράσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Για το λόγο αυτό διεξάγουμε αυτή τη στιγμή μια έρευνα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς για να έχουμε μια συνολική εικόνα για τις διαφορετικές δράσεις που χρειάζονται για να ενισχυθεί η υλοποίηση και η επιβολή της συγκεκριμένης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα. Η έρευνα αυτή θα δώσει και στοιχεία αναλυτικά για τις βέλτιστες επιλογές ε, της ε, εκπλήρωσης των υποχρέωσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα είναι έτοιμα τον Οκτώβριο φέτος. Ε, in parallel, we are also making an Ταυτόχρονα, κάνουμε αποτίμηση της, του οικονομικού, δημοσιονομικού και κοινωνικού ωφέλους που θα έχουμε από την καλή υλοποίηση της νομοθεσίας περί αποκλήτων Συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων εδώ όπου έχει φανεί να υπάρχουν ωφέλη στην πράξη και όλη αυτή η διαδικασία αξιολόγηση θα είναι διαθέσιμη πλέον για να τη συμβουλευτεί κανεί από τον Οκτώβριο. Τέλο, να φέρω ένα εγχείρημα το οποίο και πάλι ε, πρόκειται να περατωθεί ε, για να ενισχυθεί άμεσα η εποπτεία και οι διαδικασίε αδειοδότηση στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την νομοθεσία αποβλήτων. Εδώ θα συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό ε, η σύνταξη καταλόγου βέλτιστων πρακτικών για τις επιθεωρήσεις και την αδειοδότηση και αυτές ενδεικτικά ήταν κάποιες από τις δράσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή για να στηρίξουμε την καλή συμμόρφωση σε σχέση με την οδηγία περί αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φλόρεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν βεβαίως ε, βρίσκεται σε δύσκολη θέση γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Θα μπορούσε να πάει και στη διπλωματική υπηρεσία διότι προσπαθεί με τρόπο διπλωματικό να ε, καταδείξει μια δύσκολη κατάσταση. Οι παλές χώρες μέλη δεν χρειάζονται ε, συμβουλές. Πρέπει απλώς να αποφασίσουν να εφαρμόσουν πράγματα που έχουμε ε, εγκρίνει εδώ και μια δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως έχει την θέληση, αλλά δεν έχει επαρκές προσωπικό. Διότι νομίζω ότι κάποια στιγμή εν τέλει πρέπει να συρθούν πριν των δικαστηρίων ορισμένε χώρε μέλη για να αποφασίσουν επιτέλου να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι πάρα πολύ μεγάλε ελλείψει παλαιών χωρών μελών που ήταν από την αρχή στην ευρωπαϊκή κοινότητα των έξι τότε έχουν οδηγήσει στο να μην σέβονται την οδηγία ούτε και νεότερε χώρε μέλη. Χαίρομαι πάντω που ο επίτροπο βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και ίσω μάλιστα όπω είπα θα έπρεπε να σύρει ενώπιον των δικαστηρίων ορισμένε χώρε μέλη ίσω εν ανάγκη και την δική μου. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε πάλι το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Σκεφτείτε αυτά που ακούσατε και δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κιόλα. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Φλόρενς. Πολύ σημαντικό αυτό που έφυξε. Πρέπει να τονιστεί. Στην απάντησή μου προσπάθησα να περιγράψω τις δράσεις που νωρίτερα είχαν αναλυθεί πριν φτάσουμε στο δικαστήριο επίσης. Η προσφυγή στο δικαστήριο προβλέπεται ιδίω για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί αποβλήτων. 20% των παραβιάσεων και προσφυγών που έχουν έρθει στα δικαστήρια αφορούν ακριβώ την νομοθεσία αποκλήτων. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο συνεπή και συνεκτικό και χαίρομαι ιδιαίτερω για την ε, επισήμανση αυτή από εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η επόμενη ερώτηση. Του Βιτόριο Πρόντι πρόκειται για τα απορρίμματα από γύψο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει. Κύριο Πυρεύσμα, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο γίνεται περισσότερα προϊόντα πρέπει να ανακυκλώνονται. Εάν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα απορρίμματα, η οδηγία στην έκδοχή της είναι σαφέστατη λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί η χρήση των απορριμμάτων για ανακύκλωση. Και αναφέρει πέντε βήματα που πρέπει να ακολουθούμε σε μία διαδικασία η οποία προετοιμάζει για την ε, ε, εκ νέου χρήση ή ανακύκλωση τέτοιων απορριμμάτων. Όμως, η ιεράρχηση αυτή στα διάφορα βήματα δεν αποτελεί απόλυτο κανόνα, είναι μία σειρά. Οπότε, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να καταλήγουν σε επιλογές που προστατεύουν όσο γίνεται περισσότερο το περιβάλλον. Παρόλο που τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν την διακριτική ευχέρεια για να αποφασίσουν με ποιο τρόπο ε, θα ε, χρησιμοποιήσουν τα απορριμματά, αν θα τα ανακυκλώσουν δηλαδή, αν θα τα χρησιμοποιήσουν αλλιώς κτλ. Υπάρχει και το άρθρο 11 της παραγράφου 2 της οδηγίας, όπου λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα βάσει στόχου μέχρι 50% των υλικών, οικοδομικών υλικών να ε, περνούν στην ανακύκλωση μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει βέβαια και για τα απορρίμματα από γύψο, αντί να καταλήγουν στις χωματερές. Για αυτήν την συγκεκριμένη λοιπόν απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα απορρίμματα από γύψο, η απόφαση του Συμβουλίου 33 του 2003 έχει να κάνει με τα κριτήρια αποδοχής απορριμμάτων γύψου στις κομματερές και λέει ότι τα υλικά αυτά μπορούν να πηγαίνουν σε χωματερές, σε ε, ειδικές ε, συσκευασίες εκεί όπου πρόκειται για χωματερές που δεν είναι ειδικά για επικίνδυνα προϊόντα και ότι δεν πρέπει να είναι πάνω από 5%. Άρα λοιπόν ε, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό της, ε, των ποσοτήτων που αποδομούνται. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία. Στο Συμβούλιο έχουν φροντίσει ε, να περάσουν και σε εθνικό επίπεδο, στην εθνική νομοθεσία. Όμως στην πράξη, έτσι όπως αναφέρει και η ερώτηση εδώ, η απόφαση του Συμβουλίου και πιο πολύ τα εφαρμοστικά μέτρα στα κράτη-μέλη παραβιάζουν την ουσία. Οι αρχές πρέπει να αναλάβουν δράση ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για αυτήν την ε, ενημέρωση. Σημειώνω όσα είπατε και με κάποια πλήψη δυστυχώς διότι εδώ ο γύψος είναι από αυτές τις ουσίες που θα μπορούσαν άμεσα να ανακτηθούν σε ό,τι αφορά την ε, τέλεια ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση δηλαδή κάποιων ε, υλικών Επιφυλάσσουμε λοιπόν για να ξαναδούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό το μέτρο, δεδομένου ότι η έλλειψη κάποιου συστήματος εδώ για το θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην εκπομπή θείου. Ιδίω με το θείο θήκοξη, το οποίο είναι πρόδρομος άλλων υπογόνων ουσιών. Θα πρέπει λοιπόν να, τηρήσει, να βρίσκεται σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπεριφορά των κρατών μελών, όχι μόνο ως προς την θεωρητική υλοποίηση των κανόνων αυτών αλλά και ω προ την πρακτική του. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τις πληροφορίες της. Ευχαριστούμε. Ευρωπαϊκή... Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευχαριστούμε για τη συμμετοχή της και σε αυτή την ερώτηση. Επόμενη ερώτηση τώρα από την κυρία Λάγκε. Ο κύριος Φλόρεντς όμως την αντιπροσωπεύει εδώ και πρόκειται για την οδηγία πλαίσιο για τα υδατά. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τον κύριο Νικόλα Κοτάου. Uh, Ευχαριστώ. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα έχει να κάνει κυρίως με την προστασία πηγών πόσιμου ύδατος. Υπάρχει ειδική διάταξη που είναι το άρθρο 7 στην οδηγία αυτή πλαίσιο, η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση εντοπισμού των ε, πηγών που χρησιμοποιούνται για το πόσιμο είδωρ. Και όταν έχουν εντοπιστεί πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο προστατευμένων περιοχών. Επ' αυτού λοιπόν τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι στο καθεστώς επεξεργασίας υδάτων το πόσιμο είδο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές έτσι όπως αυτές προβλέπονται από την οδηγία. Γι' αυτό μιλάμε και για προστατευμένες περιοχές όπου βρίσκονται οι πηγές από τις οποίες ε, παίρνουμε το πόσιμο είδο. Ο τελικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να, να μειώσουμε τα ποσοστά επεξεργασίας στα οποία υποβάλλεται το πόσιμο είδωρο. Τα κράτη-μέλη μπορούν να λαμβάνουν διάφορα μέτρα υπάρχει ελαστικότητα δηλαδή σε αυτό από την οδηγία. Μεταξύ άλλων αναφέρεται λοιπόν και ο καθορισμός και η προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2010 τα δικά του σχέδια διαχείρισης που χρησιμοποιούνται στην οδηγία αυτή. Η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια αυτά και θα ετοιμάσει τον Εύριο του 2012 έκθεση στην οποία θα αναφέρει τα συμπεράσματά της από την αξιολόγηση αυτή όσον αφορά τις προστατευμένες περιοχές για το πόσιμο είδωρο. Τώρα το δεύτερο τμήμα της ερώτησης έχει να κάνει πιο συγκεκριμένα με την δυνατότητα χρήσης της κοινή γεωργικής πολιτικής και κυρίως της μεταρρύθμισής της για να αποζημιωθούν οι αγρότες εκείνοι οι οποίοι χρειάζεται να επενδύσουν για να προσαρμοστούν στους στόχους της οδηγίας αυτής. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι η πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου, που είναι ο δεύτερος πυλώνας της κοινή ζωικής πολιτικής, προβλέπει δυνατότητα οικονομικών ενισχύσεων για αυτή την περίπτωση. Γίνεται λοιπόν αυτό μέσω του άρθρου 38 του κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και μέσω περιβαλλοντικών μέτρων που είναι το άρθρο 39 του κανονισμού αυτού. Φυσικά και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών μέσω της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τέλος, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που υιοθετήθηκε στα τέλη του 2010 συμπεριλαμβάνονται προτάσεις και ιδέες για το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ και αναφέρονται εκεί και μέτρα που έχουν να κάνουν με οικολογική αγρανάπαυση κλπ. κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζονται. Τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με αυτά που περιλαμβάνει η, η συγκεκριμένη οδηγία για την πολλαπλή συμμόρφωση. Είναι πράγματα το οποία θα συμφωνηθούν στην Επιτροπή όταν θα έχουμε συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις. Υπενθυμίζω πάντως ότι η οδηγία για τα ύδατα Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στη Βουδαπέστη υπό την Ουγγρική Προεδρία το Μάιο, οι διάφορες εθνικές αρχές είπαν ότι θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση και ότι πρέπει να σας πω ότι τα ίδια έχουν πει και οι αρμόδιοι συγητές από την ε, ΟΚΕ, για παράδειγμα, ή και την Επιτροπή των Περιφερειών επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Φλόρενς. Η Κομισιόν μίλησε πολύ για εφαρμογή κλπ, αλλά δεν απάντησε το ερώτημα. Η ερώτηση είναι όταν επιβάλλει η Ευρώπη χώρους, περιοχές προστασίας των νερών και στόχους. Το ερώτημα είναι τότε τι γίνεται με τους γεωργούς οι οποίοι υφίστανται τότε σημαντικούς περιορισμούς απέναντι στους γείτονές τους οι οποίοι βρίσκονται σε ζώνες άλλες ε, εκτός προστασίας νερών. Άρα μπορούμε να επιβάλλουμε κανονισμούς, το ερώτημα όμως που τίθεται είναι με ποιον τρόπο αντισταθμίζονται οι ε, περιορισμοί. Οι γεωργοί δεν ζητούν περισσότερα χρήματα, αλλά επιστροφή των ζημιών. Οι παράγραφοι 38 και 39 δεν ε, θέτει το ερώτημα εάν πρέπει να δοθεί αποζημίωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Φλόρεντ λοιπόν έθεσε μια ερώτηση και θα ήθελε μια απάντηση. Εσείς κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ. Όταν μιλούμε για εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου θα πρέπει να εξετάσουμε δύο στοιχεία. Πρώτο, το γεγονός ότι η οδηγία είναι οδηγία πλαίσιο προβλέπει λοιπόν ορισμένες υποχρεώσεις που οφείλουν ε, να εφαρμόζουν οι χώρες μέλη και μετά συγκεκριμένα μέτρα στο επίπεδο του συγκεκριμένου αγροκτήματος. Τα μέτρα αυτά, ορισμένα εκ των μέτρων αυτών, είναι αμοιβαίω επωφελή. Δηλαδή δεν επιβάλλουν πρόσθετο κόστος σε βάρος των γεωργών και ιδίω εφόσον το κόστος αυτό κριθεί ε, μέσω και μακροπρόθεσμα. Τα μέτρα, για παράδειγμα, για την ποσότητα των νερών και για την αποτελεσματικότητα χρήσης τους ε, θα έχουν σχέση, για παράδειγμα, με την εξοικονόμηση νερού από την εκμετάλλευση και επομένως θα πληρώνουν και λιγότερα και θα διατηρούν το νερό για χρήση στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν ένα στοιχείο κόστους και ωφέλους που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα, για τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού ανάπτυξης της υπαίθρου προσφέρουν την δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας και για την ποσότητα και για την ποιότητα. Είναι σαφές ότι εξετάζουμε εδώ την σχέση μεταξύ WFT και αυτό για την πολλαπλή συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή βέβαια θα πρέπει να αναθεωρηθεί η διάταξη που μόλις ανέφερα. Σας ευχαριστώ κύριε Φλόρεντς. Ίσως ο κύριος Φλόρεντς να έχει διαφορετική άποψη σχετικά με το κόστος το οποίο εν τέλει επομίζονται οι Γεωργοί. Αλλά εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και προχωρούμε στο τελευταίο θέμα του κυρίου Κριστέιβης για την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η κυρία Σίλβια Άρελεϊ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει τα σημεία όπου μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στη συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χώρων μελών για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, του δικαίου της Ένωσης δηλαδή. Ένα από τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι η απέτηση να συνοδεύεται κάθε νέο νομοθέτημα από ένα σχέδιο επιβολής για την οδηγία για την 2007-60 και σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες οδηγίες χρήσης των ζώων και ε, βιομηχανικών αποβλήτων. Αυτά τα λεγόμενα checklist της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ε, παρακολουθούνται από τους ειδικού της χώρες μέλη. Και σε ό,τι αφορά την οδηγία χρήσης των ζώων, εμείς καταστήσαμε διαθέσιμο ένα υπόμνημα για την μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των βασικών διατάξεων για να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να μεταφέρουν δηλαδή στο δίκαιό τους τις ε, οδηγίες και για την εφαρμογή επίσης και αυτό το checklist δημιουργήθηκε μαζί με συνεργασία των εμπειρογνωμόνων των χωρών μελών. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος πρότεινε επίσης τις χώρες μέλη και ιδιαίτερα για την οδηγία χρήσης των ζώων να δημιουργηθούν ομάδες ε, στο εθνικό επίπεδο που θα παρακολουθούν τις, τους συγκεκριμένους φακέλους, τα συγκεκριμένα ντοσιέ με συμμετοχή εθνικών εμπειρογνώμων και στο τοπικό και στο περιφερειακό επίπεδο με συγκεκριμένα καθήκοντα επιβολής ώστε οι χώρες μέλη να εμπλέξουν τους τοπικούς τους αξιωμα, αξιωματούχους με τον ίδιο τρόπο που προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εμπλέξει εθνικούς αξιωματούχους στην ε, εφαρμογή. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρακολουθεί την έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ε, διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 275 της Συνθήκης και με την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ε, συνθήκης. Τρίτο, προβαίνουμε και σε αξιολόγηση της ε, συμμόρφωσης των μέτρων μεταφοράς όσο είναι το δυνατόν περισσότερο. Τέταρτο, αναπτύσσουμε κατευθυντήριες γραμμές για να υποστηρίξουμε τις εθνικές αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και τους ε, διαφόρους άλλους ενδιαφερομένους για παράδειγμα ε, στον τομέα των απορριμμάτων έχουμε δημοσιεύσει έγγραφα στην ιστοσελίδα μας με συνήθως υποβαλόμενες ερωτήσεις και ούτω καθεξής. Επίσης αναφέρω πρόσφατες μελέτες για την εφαρμογή και για την επιβολή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και αργότερα φέτος θα εγκριθεί σχετική ανακοίνωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά το τελικό της περιεχόμενο ακόμα δεν είναι γνωστό πάντως θα είναι knowledge based και θα αναφέρεται επίσης και σε θέματα εκπομπής ε, ε, αερίων θερμοκηπίου. Και στις 15 Ιουνίου 2011, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε διάσκεψη των ενδιαφέρων μερών με συζήτηση δύο θεμάτων, βελτίωση δηλαδή της βάσης γνώσεων, ήδη πόροι, συνεργασία δικτύων, νομικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις περιβάλλοντος. Αυτά προσέφεραν, πολλαπλή, προσέφεραν γνώσεις πολλαπλούς προσέγγισης και τεχνικών με χρήση σχετικών στατιστικών για την ε, χρήση των ιδίων πόρων, για την δημιουργία ικανοτήτων, τη συνεργασία μεταξύ ομάδων εμπειρογνωμόνων και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο την ε, δυνατότητα να υποβάλλονται καταγγελίες και άλλα θέματα. Με συμμετοχή πολλών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, άλλα δίκτυα, την Ιντερπόλ, πανεπιστημιακούς, επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, μη κρατικών οργανώσεων και ιδίως της ε, περιβαλλοντικής ε, οργάνωσης, η Ουγγρική Προεδρία καθώς και η επόμενη Πολωνική Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε. Είναι τα τελευταία λεπτά της συνεδρίασής μας. Ο κύριος Ντεβίς οπωσδήποτε θέλει να θέσει ερώτηση. Oh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξέπληξε που έδωσε τόσο διεξοδική απάντηση. Δεν μπορούσαμε να σας κάνουμε να σταματήσετε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερω. Κατά πρώτον, μπορούσατε την απάντηση αυτή να τη διαθέσετε και τον Πρόεδρο για να τη μοιράσει στα μέλη τη Επιτροπή. Ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική. Και δεν θέλω εδώ να δώσω μεγάλη συνέχεια, αλλά σε σχέση με την πρώτη σας παρατήρηση για τα κοινά προγράμματα και τις κοινούς καταλόγους ελέγχου ξέρουμε ότι είναι δύσκολο τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις για τους πίνακες συσχετισμού. Όταν λοιπόν λαμβάνει τέτοιες δράσεις η Επιτροπή τι είδους ε, αντίδραση περιμένει κάτι τα μελη είναι δεσμευτική απέτηση. Ναι. Πώς το καλύπτεται αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να σας επισημάνω ότι έχουμε δημοσιεύσει και όλες τις πληροφορίες και για την διάσκεψη και τις παρουσιάσεις και ό,τι αφορά την περιβαλλοντική μας πολιτική στην, στον τόπο της Europa. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα, μπορείτε να τα κοιτάξετε. Να θυμίσω ότι η διάσκεψη θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο. Και για τους πίνακες συσχετισμού που ρωτήσατε, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος μετά την περίοδο μεταφοράς και τη λήξη της θα ασχολείται συστηματικά και διαρκώς με την αποτίμηση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας των κρατών μελών. Αυτό θα γίνει ταυτόχρονα για όλα τα κράτη-μέλη. Θα υπάρξει πλήρως ισότιμη μεταχείριση. Και θα έχουμε συνεκτική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί και συμβούλους από τις υπηρεσίες μας εσωτερικώς για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τους πίνακες συσχετισμού. Αυτά είχα να πω για το θέμα αυτό. Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, ε, μπορείτε την αρχική απάντηση να μας τη μοιράσετε. Θα υπάρξει αντίγραφο, σας παρακαλώ. Ναι, παρακαλούμε αν μπορείτε στην Προεδρία να προωθήσετε την παρουσίασή σας, ώστε να την φωτοτυπήσουμε και να τη μοιράσουμε στους βουλευτές. Σας ευχαριστούμε κυρία Άιντερ. Φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Το σημείο 8 τα της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής ΕΝΒΗ στην ε, Πολωνία θα το δούμε στις 3 μετά την εξέταση του σημείου 9 τις βιωσιμότερες γεωργικές πρακτικές, αλληλευτικές μάλλον πρακτικές στην Βαλτική, την ακρόαση ακριβώ που θα λάβει η χώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Merci.